Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, καθίστε παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε για να μην μας ξεφύγει και ο χρόνος. Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο συνεδρίες. Τη συνεδρία υπεριθμών 3 αυτού του διήμερου σεμιναρίου για την προστασία των δεδομένων και για τις προκλήσεις ε, στην επιβολή του νόμου. Και έχουμε και τη συνεδρία υπαριθμών 4 για αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για επεξεργασία δεδομένων και αυτούς που επεξεργάζονται τα δεδομένα στον ιδιωτικό τομέα και στον τομέα τη απασχόληση. Πριν ξεκινήσουμε όμως τι συζητήσει, τις οποίες θα συντονίσουν ο κύριος Δημήτριος Δρούτσα και ο κύριο Σον Κέλλη, αντιστοίχω την Τρίτη και την Τέταρτη, έχουμε την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ, που είναι η Επίτροπος υπεύθυνη για το σημαντικό χαρτοφυλάκιο των δικαιωμάτων και της ε, δικαιοσύνης. Και γι' αυτό είναι η βασική Επίτροπος μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, ασχολείται με αυτή την πρωτοβουλία για την προστασία δεδομένων για την πρόταση κανονισμού και για την πρόταση οδηγίας για την προστασία δεδομένων. Αυτά τα οποία συζητήσαμε και σήμερα το πρωί και που θα συζητήσουμε και σήμερα το απόγευμα και αύριο όλη μέρα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ, και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Σας προτείνω λοιπόν Όσοι θέλετε να λάβετε το λόγο παρουσία της Επιτρόπου, να σηκώνετε το χέρι σας για να σας καταγράφουμε. Και μετά την παρουσίαση της κυρίας Ρέντινγκ, θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Κυρία Ρέντινγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι με εντυπωσίασε η ημερήσια διάταξη την οποία έχει προετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια ημερήσια διάταξη που μας δίνει πραγματικά τροφή για εργασία και συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και στα οποία πρέπει να συνεισφέρουν όλοι οι αιρετοί που έχουν την ευθύνη για τα δικαιώματα των πολιτών αφενός και για την σωστή λειτουργία της οικονομίας αφετέρου, διότι θέλουμε να συνδυάσουμε αυτά τα συμφέροντα και σε αυτό θα συνεισφέρουν οι εκπρόσωποι και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί την αρχή μιας νέας φάσης για την προστασία δεδομένων και τα θέματα που έχετε επιλέξει για τις συζητήσεις σας βρίσκονται στην καρδιά του θέματος της προστασίας δεδομένων. Μιλάτε για τις βασικές αρχές, προστασία ε, του ατόμου, ανάπτυξη της οικονομίας, επιβολή του νόμου και σχετικές προκλήσεις. η διακυβέρνηση που θα οδηγήσει σε συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία και πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να βρούμε τις σωστές απαντήσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει για τις συζητήσεις αυτές έχει επιλεγεί εξαιρετικά, διότι η δημιουργία εμπιστοσύνης μέσα στον παγκόσμιο χώρο είναι στον πυρήνα αυτών που πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζετε ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων ξεκινούν από το 1995. Μόνο το 1% του πληθυσμού είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο τότε. Μιλάμε για την εποχή πριν από το διαδίκτυο και ο δημιουργός του Facebook ε, ήταν 8 χρονών. Δεν υπήρχαν ε, σύννεφα αποθήκευσης δεδομένων. Τα σύννεφα ήταν αυτά τα οποία πάντοτε γνωρίζαμε στην ατμόσφαιρα. Ξεκίνησε μια καινούργια οικονομία όμως με το διαδίκτυο και τα προσωπικά δεδομένα έχουν γίνει πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία και υπάρχει μια τεράστια αγορά. Αναπτύσσεται κατά 40% ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δεδομένα λοιπόν αποτελούν ένα νόμισμα ανταλλαγής σε αυτή τη νέα ψηφιακή οικονομία. Και όπως οποιοδήποτε άλλο νόμισμα για να μπορέσει να είναι επιτυχημένο πρέπει να έχει και δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας και η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό. Δημιουργούμε ενιαίους κανόνες για όλη την εσωτερική αγορά και επίσης γνωρίζετε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία οποιοδήποτε νομίσματος εξαρτάται από ένα πολύτιμο εμπόρευμα και αυτό το πολύτιμο αγαθό είναι η εμπιστοσύνη και μόνο όταν υπάρχει προστασία του καταναλωτού, τότε θα προστατεύονται, ότι όταν υπάρχει προστασία των ε, καταναλωτών και υπάρχει εμπιστοσύνη από τους καταναλωτές ότι θα προστατεύονται τα δεδομένα, τότε θα τα εμπιστεύονται ώστε να μπορούν να τα ε, χρησιμοποιούν ως νόμισμα στην ε, ψηφιακή οικονομία. Το 70% των πολιτών μας πιστεύουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που χρησιμοποιούν οι εταιρείε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και όχι για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συνελέγησαν. Εάν ε, δεν μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση, αν δεν έχουμε κανόνες αξιόπιστους που θα εφαρμόζονται με συνέπεια και που θα κάνουν ε, τα δεδομένα πιο εύκολα και, πιο, και λιγότερα δαπανηρά στη χρήση τους και θα εμπνέουν και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τότε θα έχουμε πραγματικό πρόβλημα, διότι η ψηφιακή εσωτερική αγορά δεν θα αναπτυχθεί στον βαθμό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία ανάπτυξης στην ε, ψηφιακή αγορά. Δείτε ε, το cloud computing. Ε, ήδη υπάρχουν σημαντικές οικονομίες και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες με αυτή την με το νέο τομέα στο πλαίσιο της, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέχρι το 2020 μιλάμε για τεράστια αγορά, πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να επιταχύνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις διαδικασίες ανάπτυξης αυτών των προϊόντων, ούτως ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί και υπάρχει ένας φραγμός ε, που ακόμη είναι παρόν, δηλαδή ο φόβος των πολιτών ότι η χρήση νέας τεχνολογίας ε, ε, κρύβει και νέους κινδύνους. Και όταν λέω πολίτες, εννοώ όλα τα άτομα που ανησυχούν για το τι συμβαίνει με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως επίσης και οι υπηρεσίες που ανησυχούν για την ασφάλεια των δεδομένων τους ή και για ενδεχόμενη ε, διαταραχή των, ε, της λειτουργίας τους ε, λόγω των δεδομένων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στα clouds στο νέο αυτό προϊόν. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε αυτό το νέο ψηφιακό τομέα, πιστεύω ότι είναι επίγον να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Συγχαίρω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που επέλεξε την προστασία δεδομένων ως θέμα για την ε, κοινοβουλευτική ε, συνάντηση αυτής της χρονιάς και χαιρετίζω το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα που τόνισαν ο κύριος Άλμπρεχτ και ο κύριος Δρούτσας, οι δύο εισηγητές ε, της ΛΥΜΠΕ. Αυτό θα μας δώσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για την μεταρρύθμιση μέχρι το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας αφού θα έχει προετοιμαστεί από την Κυπριακή Προεδρία. Περιμένω και το σχέδιο έκθεσης κατά τους επόμενους μήνες και έτσι οι συζητήσεις μας θα επιταχυνθούν. Σας διαβεβαιώνω ότι θα έχετε την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής που θέλει να προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Θα δώσουμε την πλήρη μας υποστήριξη και στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε να έχουμε κανόνες που θα είναι κατάλληλοι για τον 21ο αιώνα. Η σημερινή μας συνάντηση είναι ιδιαίτερα εύστοχη και ε, βλέπω ότι υπάρχουν και πολλά ερωτήματα τα οποία τέθησαν για να απαντηθούν γραπτός, δεν απαντήθηκαν όλα γραπτός, αλλά για να κάνω την εισαγωγή των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν θα ήθελα ε, να δούμε τα σημεία αυτά τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Εσείς ως Εθνικά Κοινοβούλια ενδιαφέρεστε για τη σχέση μεταξύ του πακέτου μεταρρύθμισης ε, και της εθνικής νομοθεσίας. Θα διαρωτάστε γιατί προτείνει ένα κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν προτείνει μια οδηγία. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρη. Προτείνουμε κανονισμό, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό μέσα στην ενιαία αγορά και είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την ε, επιβολή ε, των νόμων προστασίας δεδομένων παντού. Η οδηγία του 95 κατέληξε σε 27 διαφορετικά και συχνά αντιφατικά συστήματα κανόνων προστασίας δεδομένων. Πολλά διαφορετικά πρότυπα που οδήγησαν σε περιτά γραφειοκρατικά εμπόδια. Και αυτό επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ακριβώς είναι αυτές που παραπονούνται εδώ και χρόνια για τις δυσκολίες που έχουν και για το κόστος το οποίο συνεπάγεται η εφαρμογή των 27 διαφορετικών κανόνων όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες στην εσωτερική αγορά. Άμεσα λοιπόν εφαρμοζόμενη νομοθεσία είναι ένας κανονισμός που θα δώσει ασφάλεια δικαίου εισάγοντας ένα εναρμονισμένο σύστημα κανόνων, δηλαδή θα δημιουργήσει μία ενιαία αγορά ανοιχτή και χωρίς φραγμούς, χωρίς εθνικά σύνορα. Επίσης γνωρίζω ότι γίνεται μία συζήτηση για την προστασία δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα και υπάρχει συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχουν διαφορές. Αυτό το οποίο υποβάλλουμε δεν είναι κάτι καινούριο ήδη στην οδηγία του 1995 δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου. Δεν έχουμε κάνει λοιπόν θεμελιώδεις αλλαγές στην νομική κατάσταση εδώ. Η διάκριση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού χώρου δεν είναι και σαφής εξάλλου. Και οι τεχνολογικές αλλαγές συγχαίουν όλο και περισσότερο το τοπίο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι γίνεται εάν ε, μια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ε, ε, ανεβάσει σε ένα υπολογιστικό νέφος δεδομένα που αφορούν μια ιδιωτική εταιρεία. Πού ξεκινά το ιδιωτικό και πού τελειώνει το δημόσιο και πού συνδυάζονται τα δύο. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους νομικούς αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό που σας εξήγησα λοιπόν σημαίνει ότι δεν δικαιολογείται καμία διαφοροποίηση. Όχι, διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει διαφοροποίηση. Οι δημόσιες αρχές κάνουν την επεξεργασία δεδομένων ε, με βάση το δημόσιο συμφέρον και όχι με βάση τη συγκατάθεση ή με βάση ε, τα άλλα θέματα. Ο κανονισμός ε, ε, επισημαίνει συγκεκριμένους τομείς όπου δικαιολογείται μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ακολουθήσει οι ίδιες αρχές. Περιορισμός του στόχου, περιορισμός των δεδομένων, ε, ιδιωτικότητα εξορισμού, εγγύηση προσωπικών δικαιωμάτων, αυτά ισχύουν και για τον δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα. Δεν μπορεί να θεωρείται ότι ε, είναι αυτονόητο ότι ο ιδιωτικός τομέας πάντοτε τα τηρεί εάν δεν υπάρχουν σαφώς ε, μέσα στην νομοθεσία. Σε αυτό το νέο τοπίο προστασία δεδομένων θα συνεχίσουν να παίζουν ένα ρόλο και τα εθνικά κοινοβούλια. Ο προτινόμενος κανονισμός ε, αναφέρει συγκεκριμένους τομείς πολύ ευαίσθητους σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι επαφίονται στο εθνικό δίκαιο, παραδείγματο χάρη. Πώς θα έχουμε ισορροπία μεταξύ προστασίας δεδομένων και ελευθερίας έκφρασης. Κατά πόσο είναι θεμητή η επεξεργασία δεδομένων. Εφόσον τηρούνται οι γενικές αρχές του κανονισμού, μπορούν οι εθνικές νομοθεσίες να προσθέτουν στοιχεία στον τομέα της ελευθερίας έκφρασης παραδείγματος χάρη. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική λύση, διότι ο κανονισμός αναγνωρίζει ότι σε ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι για τα κράτη-μέλη, πρέπει να αφήνουμε Αντίστοιχε αρμοδιότητε στα κράτη-μέλη. Τα Εθνικά Κοινοβούλια θέτουν ερωτήσεις και για το ρόλο της Επιτροπής και των ε, Εθνικών Αρχών. Όσον αφορά το ρόλο της Επιτροπής, γνωρίζω ότι έχουν εκφραστεί πολλές ανησυχίες για τον ε, αριθμό, για το πόσες ε, εξουσίες θα έχει η Επιτροπή, για το αν θα αποφασίζει να εκδίδει πράξεις κατά εξουσιοδότηση ή εφαρμοστικές διατάξεις. Θελήσαμε να κάνουμε την νομοθεσία αυτή τεχνολογικά ουδέτερη. Αυτό ήταν ηθελημένο, διότι το να προκύψει ένας κανονισμός είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία και δεν μπορούμε να αλλάζουμε τον κανονισμό κάθε φορά που αλλάζει η τεχνολογία. Θέλουμε λοιπόν οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, να υπάρχουν και να τις ακολουθούμε, να μην τις εμποδίζουμε. Επομένως, ο κανονισμός έπρεπε να είναι ε, ευέλικτος, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογία που αλλάζει και τις ε, καταναλωτικές πρακτικές που αλλάζουν. Και γι' αυτό υπάρχει η διάκριση μεταξύ πράξεων κατεξιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Θέλουμε οι κανόνες και οι διατάξεις του κανονισμού να ισχύουν για τις τεχνολογικές εξελίξεις του μέλλοντος, ε, χωρίς να χρειάζεται μια πλήρης μεταρρύθμιση του κανονισμού και η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν πράξεις κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις ακριβώς για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Τούτου λεχθέντος δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει διαφωνία επί της αρχής της χρήσης πράξεων κατεξουσιοδότηση. Αλλά για τους ε, διάφορους τύπους πράξεων κατεξουσιοδότηση μπορεί να γίνει σχετική συζήτηση και ευχαρίστως να εξετάσουμε το πεδίο και τον αριθμό των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, εάν οι νομοθέτες αυτό το θεωρούν σημαντικό. Εάν θεωρείται σημαντικό να περιορίσουμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση μόνο στην περίπτωση που έχουμε που θέλουμε να έχουμε ευελιξία για τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την γνώμη σας ε, για τις δυνατότητες της Επιτροπής, για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και να μου προτείνετε και εναλλακτικέ λύσεις κατά τη γνώμη σας. Για να σας βοηθήσω σε αυτή τη διαδικασία προβληματισμού, το να μπουν λεπτομέρειες σε μια νομοθετική πράξη σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ευελιξία και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Το να αφήσουμε υπερβολικά στοιχεία προς ρύθμιση στα κράτη-μέλη μας απομακρύνει από το στόχο του να έχουμε ένα δίκαιο πεδίο, σε μια, δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού σε μια ανοιχτή αγορά. Τρίτον, αν είχαμε προσεγγίσει συγκεκριμένες ανατομέα θα γίνει πιο πολύπλοκο το νομοθετικό περιβάλλον και όχι απλουστευμένο όπως θα το θέλαμε. Και τέταρτον, κώδικας είναι κάτι που πολύ συχνά δεν θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Βέβαια, όπως σας είπα, είμαι και πρόθυμη να εξετάσουμε κάθε πράξη καταξουσιοδότηση μία προς μία, να δούμε κατά πόσο είναι απαραίτητη η κάθε πράξη καταξιοδότηση ή μήπως μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Ένα δεύτερο στοιχείο τώρα. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων. Οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων θα παραμείνουν η ραχοκοκαλιά της επιβολής των κανόνων προστασίας δεδομένων. Αυτό είναι δική μας επιλογή, διότι σε ε, μία στη λογική μιας ενιαίας αγοράς θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιλογή να έχουμε μία κεντρική αρχή προστασίας δεδομένων για όλη την ενιαία αγορά. Αλλά εγώ επέλεξα να μην το κάνουμε έτσι. Επέλεξα να έχουν την ευθύνη οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων που θα προσπαθήσουν να οργανώσουν τη δουλειά τους ε, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα από τις εθνικές αρχές και αυτό θα ενισχύσει τη βαρύτητα της νόμης τους, θα εξασφαλίσει μια εναρμονισμένη διαδικασία για θέματα που έχουν ευρωπαϊκή σημασία είτε για γενικότερα θέματα προστασίας δεδομένων, είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις και οι αρχές προστασίας δεδομένων θα αλληλοϊποστηρίζονται και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν και η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτήμους λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία 1.500 υπευθύνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα δώσει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα στις αρχές προστασίας δεδομένων κάθε φορά που θα θέλουν να είναι αντιμέτωπες με τις εθνικές κυβερνήσεις ή με την Επιτροπή ή με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο ρόλος της Επιτροπής σε αυτό το μηχανισμό συνεκτικότητας είναι πολύ σαφής. Είναι το σημείο τελευταίας προσφυγής, δηλαδή η Επιτροπή βρίσκεται εκεί μόνο για λόγους ε, ασφαλείας. Θα χρειαστεί ο ρόλος της Επιτροπής μόνο εάν αυτά τα οποία αποφάσισαν οι εθνικές αρχές υπάρχει αμφιβολία αν είναι συμβατά με την εθνική νομοθεσία ή αν υπάρχει κίνδυνος μη συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων. Και δεν εφευρίσκω κάτι νέο εδώ, διότι ο μηχανισμός αυτός υπάρχει και σε άλλους ε, τομείς, όπως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και έχει λειτουργήσει πολύ σωστά. Η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να γίνει μια υπερ-αρχή προστασίας δεδομένων. Ούτε είναι δουλειά μας, ούτε θα είναι δουλειά μας στο μέλλον και δεν μπορεί και να είναι δουλειά μας. Οι αρχές προστασίας δεδομένων πρέπει να προσδιορίζουν το τι θα γίνεται σε κάθε περίπτωση και όχι η Επιτροπή. Μόνο εάν σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις τίθενται γενικότερα ζητήματα, ίσως χρειαστεί ως τελευταία προσφυγή να καταλήξουμε στην Επιτροπή ως διαιτητή. Αλλά αυτό θα είναι μόνο κατεξαίρεση και δεν θα συμβαίνει ως γενικός κανόνας. Άλλη σημαντική ερώτηση που τίθεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν θα είναι κανονισμός ή οδηγία. και εγώ, αλλά πιστεύω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύουμε ότι το αν θα είναι κανονισμός ή οδηγία θα πρέπει να το δούμε ως πακέτο. Η ελευθερία και η ασφάλεια των πολιτών είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Είναι δύο στόχοι πολιτικής, τους οποίους πρέπει να επιτύχουμε με την υιοθέτηση των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων. Μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκομένους και με τις αρχές των κρατών μελών, καταλάβαμε ότι οι κανόνες όπως έχουν τώρα στην απόφαση πλαίσιο δεν είναι ικανοποιητικοί. Υπάρχουν πολλοί κανόνες, διάφορα νομικά εργαλεία. Και αυτό δεν μπορεί να διευκολύνει την ε, ομαλή και απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Εδώ βασιζόμαστε στην απόφαση πλαίσιο του 2008 που θα αντικατασταθεί από την οδηγία και αυτό καλύπτει μόνο τη διασυνοριακή επεξεργασία. Και εδώ έχουμε άλλη μία από τις ερωτήσεις σας. Γιατί πρόσθεσα την εσωτερική επικοινωνία στη διασυνοριακή επικοινωνία. Μετά από μακρές συζητήσεις με αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά στην πράξη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έχουν δίκιο, διότι οι αρχές επιβολής του νόμου μας είπαν ότι δεν κάνουν τη διάκριση μεταξύ διασυνοριακής επεξεργασίας και εγχώριας επεξεργασίας των δεδομένων και δεν είναι προβλέψιμο εξ αρχής ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει ένας κράτος μέλος μπορεί να είναι αντικείμενο διασυνοριακής ανταλλαγής ή όχι. Μόνο στην πράξη, στην πραγματική δουλειά των ε, ε, αρχών ε, ασφαλείας προκύπτουν αυτά τα θέματα και δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση στην καθημερινή τους δουλειά. Παραδείγματος χάρη, μία βάση δεδομένων εθνική που χρησιμοποιείται από τις διοκτικές αρχές μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί σε εθνικό επίπεδο καθώς και προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί από ένα άλλο κράτος μέλος. Δεν θα ήταν αποτελεσματικό το να δημιουργήσουμε δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων για αυτά τα δεδομένα διότι θέλουμε να τα έχουμε μαζί. Και δεν θα ήταν και αποτελεσματικό να εφαρμόζουμε δύο είδη κανόνων προστασίας δεδομένων σε δεδομένα που υπάρχουν σε μία βάση δεδομένων. Η διάκριση είναι τεχνητή μεταξύ δεδομένων που έχουν συλλεγεί σε εγχώριο επίπεδο και διασυνοριακά. Και για θέματα επιβολής του νόμου, ένας ύποπτος για εγκληματικές ενέργειες μπορεί να είναι κάποιος εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης ή που τα στοιχεία του βρίσκονται στο σύστημα ΕΚΡΙΣ. Και αν υπάρχουν εθνικά δεδομένα, γίνονται απευθείας διασυνοριακά δεδομένα αυτά και ο αστυνομικός που τα χειρίζεται δεν γνωρίζει καν αν είναι εθνικά δεδομένα ή διασυνοριακά. Ακούσαμε λοιπόν όσα μας είπαν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές και γι' αυτό δεν κάναμε τη διάκριση μεταξύ αυτών των δεδομένων. Και το σκεπτικό είναι το ίδιο σκεπτικό που υπάρχει σε όλο τον κανονισμό και την οδηγία, δηλαδή η απλούστευση. Θέλουμε να υπάρχει απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και να είναι πιο εύκολη η συνεργασία για την επιβολή του νόμου. Ορισμένα εθνικά κοινοβούλια έχουν ε, αναφέρει την ανάγκη να δημιουργηθούν ε, συμφωνίες πριν τεθεί σε ισχύ η σχεδιαζόμενη οδηγία. Και διερωτώνται κατά πόσον αυτές οι συμφωνίες θα είναι συμβατές με τη μελλοντική οδηγία ή όχι. Η συνθήκη ως προς το θέμα αυτό είναι πολύ σαφής. Τα κράτη-μέλη νομικώς δεσμεύονται να διασφαλίσουν τη συμβατότητα των διμερών συμφωνιών τους με τις ίδιες τις συνθήκες, με, με το δίκαιο της Ένωσης και παραθέτω εδώ ε, υποχρεώνται να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξαλείψουν κάθε ασυμβατότητα που μπορεί να προκληθεί. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να λάβουμε υπόψη την νομική αυτή διάσταση. Όμως πώς αυτό μπορεί να τεθεί στην, στην σε εφαρμογή. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών ε, και να εφαρμόζονται σωστά οι συνθήκες, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κανόνες για τη μεταφορά των δεδομένων ε, διαφορετικοί από 100 μέλος σε 100 μέλους, για τη μεταφορά δεδομένων προς τις χώρες. Τα πιο προστατευτικά κράτη-μέλη μπορεί να μην μεταφέρουν τα δεδομένα σε κράτη-μέλη που δεν είναι τόσο προστατευτικά. Μπορεί να μην γίνουν αποδεκτές όλες οι διευθυντήσει στον τομέα της αποστολής δεδομένων. Μπορεί κάποιος να επικαλεστεί λόγους ασφάλειας. Καταλαβαίνω ότι η αναθεώρηση των ε, υπαρξών συμφωνιών και αναγκαία είναι, αλλά προκαλεί και διοικητικό άχθος. Γι' αυτό λοιπόν η οδηγία προβλέπει μια πενταετή περίοδο για την πρώτη αναθεώρηση. Πολύ μεγαλύτερη από ότι η διετία που προβλέπεται για την υλοποίηση της οδηγίας. Επίσης αφήνει το περιθώριο για την ε, μεταφορά, τη μεταφορά που πρέπει να γίνει αυτομάτως εάν λόγου χάρη πρέπει να αποφευθεί μια σοβαρή απειλή για την δημόσια ασφάλεια ή να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα αμέσως. Ειδικέ επιχειρησιακέ ανάγκες πρέπει να μπορούν να καλυφθούν και στο μέλλον. Ο πρόεδρος φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αγχώνεται, γιατί κοιτάζει και το πρόγραμμα. Θα σταματήσω εδώ, πρόεδρε, και θα απαντήσω στις ερωτήσεις και για τα υπόλοιπα σημεία, τα οποία δεν πρόλαβα να αναπτύξω. Thank you, Ευχαριστώ, Επίτροπε Ρέντινγκ. Έχετε δίκιο. Το πρωί καταφέραμε να κρατήσουμε το χρόνο. Ήμασταν πολύ συνεπεί και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και τώρα το απόγευμα. Έχουμε δύο γύρου συζήτηση. Και θα έχουμε και διάλογο, αλλά για την ώρα έχουμε λάβει έξι αιτήσει ε, για, από συμμετέχοντες που θέλουν το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν και προκειμένου να παραμείνουμε πιστοί στο χρονοδιάγραμμά μας, δύο λεπτά για τον καθένα. Προσπαθείτε παρακαλώ να αναπτύξετε τις απόψεις σε δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα από τη Σουηδική Βουλή ο κύριος Μπόλιν. Ο κύριος Μπόλιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά. Ήθελα να σχολιάσω την οδηγία. Ο κανονισμός, όπως είπατε, εμπνέεται από την απόφαση πλαίσιο του 2008. Απόφαση πλαίσιο που διαθετεί την ε, διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της αστυνομική και δικαστικής συνεργασίας, διασυνοριακά. Το σχέδιο οδηγία τώρα, σε σύγκριση με την ε, ισχύουσα οδηγία, προβλέπει και την εσωτερική επεξεργασία δεδομένων. Στο Σουηδικό τώρα Κοινοβούλιο, στο Σουηδική Βουλή, έχουμε την εντύπωση ότι εδώ ίσως να υπάρχει αντίφαση με την αρχή της επικουρικότητας. Και αυτό γιατί για σκοπούς δίωξης εγκληματικών ε, πράξεων εκεί που χρειάζεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών αρχών, εκεί συνήθως εφαρμόζεται η αρχή της επικορικότητας. Ιδαλώς μπορεί να υπάρξει και ασυμβατότητα με την εθνική ποινική νομοθεσία, το εθνικό ποινικό δίκαιο. Η απόφαση πλαίσιο έπρεπε να έχει μεταφερθεί πλήρως σε όλα τα κατημέρια από το Δεκέμβριο του 2010 Εδώ πιστεύουμε ότι είναι πολύ νωρί για να έχουμε ήδη διεξαγάγει συμπεράσματα και οριστικά πορίσματα για το τι έχει πετύχει η απόφαση πλαίσιο αυτό, για αν ήταν επιτυχημένη ή όχι. Θέλαμε λοιπόν και τι δικέ σα απόψει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Και τώρα από τη γερμανική Bundestag, ο κύριο Ράιχενμπαχ. Ähm, ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τους στόχους που επιδιώκεται μέσω του κανονισμού αυτού. Θέλουμε ακριβώ να έχουμε ένα κανονισμό που να επιτρέπει να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο εναρμόνιση για τόσο σημαντικά ζητήματα. Ξέρετε ότι το συνταγματικό δικαστήριο μα είπε ήδη και αποφάνθηκε ότι εφόσον πρόκειται για εθνική προστασία, ε, μπορεί να πληγεί ταυτόχρονα με την εθνική προστασία ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έχω τώρα δύο ερωτήσει να σα θέσω. Υπάρχει άμεσο σχετισμό μεταξύ των όσων προβλέπονται από τον κανονισμό για την προστασία γενικώ και την οδηγία για την ανταλλαγή δεδομένων σε τομεί αστυνομική και δικαστική συνεργασία ή πρόκειται να υλοποιηθούν ε, τα δύο αυτά νομοθετήματα με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Και έπειτα μιλήσατε και για το εθνικό επίπεδο, του εθνικού ελεγκτέ. Εδώ έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Εννοείται ότι στα πλαίσια συνεργασίας που έχουμε συνάψει με τις Ηνωμένες και άλλες τρίτες χώρες, τα δεδομένα που έχουν συγγεί λόγω χάρη στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες, δεν θα μπορούν να είναι αντικείμενο επεξεργασία και στις ΗΠΑ. Και ένα τρίτο ερώτημα. Εδώ ε, νομίζω θα πρέπει να υπάρχει σαφής συγκατάθεση, όχι για καθένα νομοθέτημα μόνον ξεχωριστά, αλλά και για την όλη διαδικασία. Ο κανονισμός στην παράγραφο 19 περιέχει κάποια στοιχεία που θέλουν να άρουν τις ε, αντιφάσεις. Δεν θα πρέπει εδώ η έννοια της συγκατάθεσης να είναι σταθερή. Διότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι υψηλό επίπεδο εναρμόνισης. Δεν θέλουμε όμως η βελτιωμένη προστασία να αποδυναμωθεί με Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέδρο Γκόμες Τελασέρνα έχει το λόγο τώρα, πρόεδρος της ε, Βουλής των Αντιπροσώπων της Ισπανίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ και για την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα προβληματισμό δικό μου, ο οποίος είναι συνάμα και ερώτηση. Και είναι ο εξή. Με τη μία... Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αμφισβητείται η δυνατότητα επέκτασης του ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα κινηθεί αυτός ο κανονισμός. Μιλώ για την πρόσβαση στα δεδομένα των, από τις υπηρεσίες ασφαλείας ενός ε, κράτους. Η γνώμη μου για το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αυτό καθεαυτό το θέμα. Το θέμα είναι η απουσία ρύθμισης σε αυτό το σχέδιο που προτείνεται. Απουσία ρύθμισης του εξής. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επαγγελματιών που δεν ανήκουν στα σώματα ασφαλείας τα κρατικά, βασικό αντικείμενο της δραστηριότητάς τους είναι η διερεύνηση, η συλλογή πληροφοριών, η απόκτηση στοιχείων ε, είτε εταιρικού χαρακτήρα, δηλαδή ε, ερευνούν άλλες επιχειρήσεις, ή ερευνούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό είναι το βασικό αντικείμενο αυτό των ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων ασφαλείας. Υπ' αυτή την έννοια, καλό θα ήταν να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να διευρύνουμε το πλαίσιο, να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο δραστηριότητας συγκεκριμένο για αυτές τις επιχειρήσεις και για αυτούς τους, επιχειρημα... τους επαγγελματίες της συλλογή πληροφοριών πιστεύουμε ότι αξίζει να εξεταστεί το εξής ενδεχόμενο, να, να δημιουργήσουμε ένα μητρό, αν όχι και ένα μηχανισμό διοικητικού ελέγχου. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, να θεσπίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια για τη δράση τους. Για τη δράση αυτών των επαγγελματιών. Π.χ το κριτήριο της αναγκαιότητας, δηλαδή μέχρι σε ποιο βαθμό είναι αδύρυτη ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένη ε, βάση δεδομένων, η αρχή του σκοπού, για ποιο σκοπό θέλουν να το κάνουν και η αρχή της αναλογικότητας, να είναι αναλογική η παρέμβασή τους με την ανάγκη που υφίσταται είναι ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την απόκτηση δεδομένων για να εξυπηρετήσει τον κόσμο των επιχειρήσεων. Δεδομένων είτε προσωπικού χαρακτήρα είτε μη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ένσιου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ρέντιν, για την παρουσίασή της. Συμφωνούμε με αυτές τις ιδέες και θέλουμε να συμπεριληφθούν σε νέα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, θέλω να τονίσω το εξής, διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων. Μιλώ για την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητων δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει μια νέα οδηγία με την οποία εναρμονίσαμε τις κυρώσεις ε, για την κατάχρηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας των πληροφοριών και το ίδιο ισχύει και για τα αδικήματα που έχουν να κάνουν με την ε, πρασία των δεδομένων, με την καταστρατήγηση δηλαδή αυτών. Αυτό όμως που μας χρειάζεται είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι βάσεις δεδομένων είναι πράγματι ασφαλείς. Πέρα δηλαδή από τις κυρώσεις σε περίπτωση ε, κατάχρησης, θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για να καταπολεμήσουμε το κυβερνοέγκλημα και τις ασφαλείς βάσεις δεδομένων. Ο κύριος Κωνσταντίν Νότς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για την εισαγωγική της παρέμβαση. Συμφωνώ απολύτως ότι η προστασία στην προστασία, η εμπιστοσύνη συγγνώμη, στην προστασία των δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρχει πρόοδος και εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και προϋποθέτηση, προϋπόθεση αυτής της ε, ε, ε, εμπιστοσύνης είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να σταματήσουν οποιαδήποτε καταχρήσεις έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια και αυτή η διαδικασία του κανονισμού πιστεύω ότι έχει πολλές δυνατότητες να προσφέρει αυτό το οποίο τελικά θέλουμε. Υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες, κανονισμός, διαδικασία. Θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να μας εξασφαλίζει την καλύτερη νομοθεσία και πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά μπορούν να προχωρούν παραλλήλως και πόσο στην κοινωνία των πολιτών αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν ε, ρόλους προστασίας των δεδομένων έχουν ε, την απαραίτητη ε, προστασία, αν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη μέσω του κανονισμού και μέσω της οδηγίας. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Θα είναι η τελευταία που θα μιλήσει από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω το εξή στην ε, κυρία Ρέντιν. Γιατί έχουμε τώρα την ε, πρόταση οδηγίας ως προς τη ρύθμιση του αριθμού των επιβατών πριν εγκριθεί το πακέτο για την προστασία των δεδομένων, πριν εγκριθεί το σχέδιο οδηγίας και το σχέδιο κανονισμού για την προστασία των ε, δεδομένων. Ξέρετε πόσο αμφιλεγόμενη είναι η πρόταση οδηγίας στην οποία αναφέρομαι. Ο ελεγκτής ε, για, τα ευρωπαϊκά δεδομέ... για την προστασία των δεδομένων ο Ευρωπαίο ελεκτή, αλλά και η ομάδα εργασίας ε, υπαριθμών 29 είπαν ότι δεν υπάρχει αναλογικότητα ούτε αναγκαιότητα ε, για αυτό το σχέδιο ε, δεδομένων. Αυτή η ομπρέλα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι μια ομπρέλα που χρησιμοποιούμε για τα πάντα και ίσω είναι υπερβολή δεν θα πρέπει να τα δεσμεύσουμε αυτά, να τα προσαρτήσουμε στις συμφωνίες που έχουμε με τις ΗΠΑ. Και πολύ συχνά ε, το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει opt-out για διάφορα άλλα θέματα και κάνει opt-in για αυτό εδώ και πιέζει όλους τους υπόλοιπους εξημών χωρίς να το έχουν συζητήσει τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι ένα εξαιρετικά ε, σημαντικό ζήτημα. Μιλούμε για ε, ευπαθή, για πολύ λεπτά δεδομένα που έχουν να κάνουν με τους επιβάτες και ε, θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες πραγματικά να ε, ε, δίνουν αναφορά για το πού κάθε το καθένας και οι συνοδοί τους και ούτω καθεξής. Είναι πλήγμα για τα προσωπικά δεδομένα. Η πλειονότητα των μελών δεν έχει υιοθετήσει νομοθεσία των κρατών μέλων για αυτό το θέμα. Δεν νομίζετε ότι πρέπει το ζήτημα αυτό να συζητηθεί εκ των προτέρων στα Εθνικά Κοινοβούλια προτού εγκριθεί η οδηγία αυτή. Ε, μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση για να εναρμονιστεί κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε κυρία Ρόμερο. Στρέφουμε προς την αξιότιμη Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς έχετε το λόγο κυρία ε, Ρέντιν. Βοηθήστε μας να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και σας παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά. Η κυρία Ρέντιν, βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε το αφεντικό. Θα μιλήσω για 10 λεπτά μόνο. Λοιπόν, δείτε τι έχουμε κάνει. Έχουμε μια οδηγία και την έχουμε φέρει προς έναν κανονισμό. Γιατί? Για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό, να έχουμε έναν κανόνα για μία ύπερο για μία ήπειρο, για τις εταιρείε μας που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και για τους πολίτες μας, ε, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι προστατεύουμε τα δεδομένα τους σε κάθε σημείο της Ευρωπαϊκής Υπήρου όπου μπορούν να υποστούν πλήγμα ή επίθεση. Δεν κάναμε το ίδιο με τη Συμφωνία Πλαίσιο. Δεν φέραμε τη Συμφωνία Πλαίσιο προς έναν κανονισμό. Γιατί? Γιατί αναγνωρίσαμε ότι μια συμφωνία πλαίσιο η οποία έχει να κάνει με πτυχές ασφάλειας, ε, πτυχές επιβολής του νόμου. Είναι μια, αυτή η συμφωνία πλαίσιο είναι επίσης ε, κάτι που άπτεται μια σειρά ζητημάτων εθνικής ευαισθησίας, μια σειρά λεπτών ζητημάτων, τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται ε, με ε, την εθνική νομοθεσία, πράγμα το οποίο γίνεται μόνο μέσω μιας οδηγίας. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος, δηλαδή ε, να προστατεύσουμε την αρχή της επικουρικότητας και να μην έρθουμε σε σύγκριση με την εθνική ποινική δικονομία και γι' αυτό το λόγο δεν επιλέξαμε την άγουσα του κανονισμού, του ευρωπαϊκού κανονισμού και επιλέξαμε την άγουσα της ευρωπαϊκής οδηγίας. Και να σας πω πάρα αυτά, ότι η νέα συνθήκη της Λισαβόνας δεν διαφοροποιεί ως προς την προστασία των δεδομένων τα δημόσιου χαρακτήρα ή προσωπικού χαρακτήρα, ιδιωτικού χαρακτήρα ε, για εμπορική χρήση ή για την πρόσβαση ε, από πλευράς αρχών επιβολής του νόμου. Η συνθήκη της Λισαβόνας εγγυάται ε, με τον ίδιο τρόπο την προστασία όλων των δεδομένων για όλους τους σκοπούς και το ίδιο προβλέπεται στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Προβλέπεται δηλαδή και μια οριζόντια προστασία. Τώρα, το επίπεδο προστασίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Τι γίνεται με αυτό, εάν το λάβαμε υπόψη μας. Δεν θα ήταν καλύτερο να διαχωρίσουμε τον κανονισμό από την οδηγία. Το κατέστησα σαφές. Ήδη, ακριβώς, χάρη ε, επειδή υπάρχει αυτή η οριζόντια προστασία από τη συνθήκη και από τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, χάρη σε αυτά δεν είναι δυνατόν σε ένα πεδίο να λάβουμε υπόψη μας τα δικαιώματα του ατόμου και σε άλλο πεδίο να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργούσε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η οδηγία και ο κανονισμός ε, αποτελούν ένα πακέτο και πρέπει να μείνουν μαζί ως πακέτο. Ναι, απαντώ ναι, προσπαθήσαμε στον κανονισμό να ε, υποβάλουμε μία πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας στις χώρες που τον προσφέρουν στα κράτη-μέλη και όχι ε, τον χαμηλότερο βαθμό προστασίας που ενδεχομένως προσφέρεται σε άλλα κράτη-μέλη. Και το κάναμε αυτό γιατί όντως πιστεύουμε ότι η προστασία των δεδομένων πρέπει να είναι ε, πράγματι ε, στεναρή. Βεβαίως το ασφαλές λιμάνι θα παραμείνει αυτή η έννοια. Ωστόσο, ως προς την επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να έχουμε πραγματική συγκατάθεση, ενημερωμένη συγκατάθεση, όχι ε, να εννοείται εμέσως η συγκατάθεση. Αυτό καθίσατε καθίσταται σαφές στον κανονισμό. Τώρα, ως προς το πολύ συγκεκριμένο ερώτημα των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας και συλλογής πληροφοριών. Πολύ συχνά ε, φαίνεται ότι στον κανονισμό δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί ξεκάθαρα η δημόσια από την ιδιωτική σφαίρα, διότι ε, το δημόσιο σκέλος συχνά αναμειγνύεται με το ιδιωτικό. Οι εισηγητές ε, έχουν ακούσει αυτό το ερώτημα επανειλημμένος ε, και αν πρέπει να ενισχυθεί ο κανονισμός για την αξιοποίηση των δεδομένων από αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σίγουρα οι συγκητές θα υποβάλουν τροπολογίες, εάν αυτό χρειαστεί. Αλλά το ερώτημα που μου ε, θέσατε εσείς ενισχύει ακριβώς ακόμα περισσότερο το επιχείρημά μου, ότι δεν πρέπει να διαφοροποιήσουμε ε, την ε, δημόσια επεξεργασία από την ιδιωτική, την, τη δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα από την ιδιωτική πρόσβαση, διότι στόχος μας είναι ε, η προστασία γενικότερα. Τώρα, θα έπρεπε να επιλέξουμε τα, προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα και σε αυτά να προσφέρουμε υψηλότερες και μεγαλύτερες εγγύησεις. Πράγματι είναι πραγματικότητα οι κυβερνοεπιθέσεις. Και πιστεύω ότι όλα τα κρατημέλη και οι εταίροι μας από άλλες υπήρους. Όλοι σταδιακά και προοδευτικά ενισχύουν τις δυνατότητες που έχουν για να καταπολεμήσουν ε, τις κυβερνοεπιθέσεις. Ωστόσο, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, αυτοί που επινοούν αυτές τις νέες μορφές εγκληματικότητας είναι ένα βήμα μπροστά από αυτούς που προσπαθούν να κάνουν την πρόληψη εναντίον αυτών των νέων μορφών ε, εγκληματικότητας. Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ανεβάσει ταχύτητα για να προσπαθούμε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Ως προς το forum shopping τώρα. Θα ήταν εσφαλμένο να συνεχίσουμε ε, με την άγουσα της οδηγίας ως προς το θέμα αυτό, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν κανόνα τον οποίο να ερμηνεύουν οι αρχές με διαφορετικό τρόπο αναλόγως ε, με την επικράτεια στην οποία βρίσκονται. Και γι' αυτό οι εθνικές νομοθετικές αρχές και ρυθμιστικές αρχές έχουν ασκήσει πίεση στο τι κάνουν οι ομόλογοι τους και δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να επιδέχεται διαφορετικών ερμηνεών ε, συγκεκριμένη, η διά, συγκεκριμένη διάταξη και εκάστοτε διάταξη, ούτως ώστε ε, δεν θέλουν να δίδεται περιθώριο για αυτό το forum shopping, να βασίζεται κάθε αρχή δηλαδή ε, σε διαφορετικό πλαίσιο για να ερμηνεύσει κατά το δοκούν. Τώρα ένα άλλο θέμα που είναι γερμανικό ζήτημα και θα το απαντήσω στα γερμανικά όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί. Δεν θέλω να σας κουράσω όλους τους άλλους με ένα θέμα που δεν το γνωρίζετε γιατί είναι περισσότερο γερμανικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί στη Γερμανία. Το ανώτατο δικαστήριο στη Γερμανία, το συνταγματικό, ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο, ε, έχει θέσει εκτός νόμου τις διατάξεις αυτές και χρειάζονται, χρειάζονται να θεσπιστούν νέες διατάξεις και η συνάδελφα Σεσίλια Μάλμστρομ που είναι υπεύθυνη στην Επιτροπή για θέματα ασφαλείας θα λάβει θέση επ' αυτού όσον αφορά την ε, περαιτέρω εξέλιξη ε, της αποθήκευσης και διατήρησης δεδομένων. Η κυρία Μάλμστρομ είναι συνεχώς σε επαφή με τον αντίστοιχο Γερμανό Υπουργό για το θέμα αυτό. Τώρα για το θέμα των δεδομένων επιβατών. Πού είναι και αυτό ένα ζήτημα προς συζήτηση. Είναι χωρίς τη συζήτηση βέβαια. Ξέρετε ότι για αυτές τις διεθνείς συμφωνίες υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει και συμβουλευτικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γνωρίζει γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των δεδομένων επιβατών, ήταν και το θέμα του SWIFT που είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Και τελικά, στο τέλος, συμφωνεί το Κοινοβούλιο με τους κανόνες αυτούς. Η συνάδελφός μου Σεσίλια Μάλστρομ και εγώ έχουμε έρθει πολλές φορές κύριε Πρόεδρε στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και έχουμε εξηγήσει τις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Πολλά υποσχόμενες όμως διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Για να αναπτύξουμε μία συμφωνία πλαίσιο με τους Αμερικανούς φίλους μας, για να μην χρειάζεται κάθε φορά να επανερχόμεθα στο θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας. Ευχαριστούμε κυρία Ρέντινγκ. Σας ακούσαμε. Μας τα είπατε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ, που ήρθατε να μας πείτε ε, τις απόψεις σας, ε, να μας παρουσιάσετε αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν δική σας πρωτοβουλία στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε. Και τώρα θα αρχίσει ο επόμενος γύρος των συζητήσεων και θα προεδρεύσει ο συνάδελφος κύριος Δημήτρης Δρούτσας. Ω συζητητής για την οδηγία για την προστασία δεδομένων και καλό και τους άλλους συμμετέχοντες στο πάνελ, τον κύριο Ντάνιελ Ντρούερ, Έλις Ντεμπούσερ, Άννα Φίλτερ και Ντιάννα Αλόνσο Μπλάς.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 Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την ε, τρίτη ενότητα των ε, εργασιών μου και ιδιαίτερα τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. And you will allow me to switch into, into English. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω στα, να συνεχίσω στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, διότι σε λίγα λεπτά θα χρειαστεί να φύγω. Ξέρω ότι δεν ήθιστε ο πρόεδρος να αποχωρεί από την ε, συνεδρίαση της οποίας πρέπει να προεδρεύει. Απλώς πολύ σύντομα να εξηγήσω, γνωρίζετε στην χώρα μου, την Ελλάδα, έχουμε μια αποφασιστική καμπή, ίσως και θετική ε, καμπή. Γνωρίζετε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η Γερμανίδα Καγκελάριος επισκέφθηκε σήμερα την Αθήνα και εγώ πολύ τελευταία στιγμή προσεκλήθη για τηλεοπτική συζήτηση σε γερμανικό κανάλι. Με συγχωρείτε λοιπόν, αναγκάστηκα να αποδεχτώ αυτή την πρόσκληση, αλλά θεώρησα σημαντικό να, ακουστεί, να μια ελληνική φωνή στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειλικρινή λοιπόν, ε, συγγνώμη, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω, αλλά ο κύριο Φως ε, έχει αναλάβει να με αντικαταστήσει, είναι σκέφτο εξηγητή για την οδηγία αυτή από την πλευρά του ΕΛΚ και είναι και συντάκτης ε, της σχετικής νομοδότησης στην Επιτροπή Γιούρι, νομικών υποθέσεων δηλαδή. Να άλλο ένα παράδειγμα τη πολύ αρμονική ελληνογερμανική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, Άξελ, για αυτή τη χάρη. Να μην σπαταλήσω τώρα άλλο χρόνο με τη δική μου την παρέμβαση. Βλέπετε ότι η προσέγγιση μας περιγράφεται αδρά στο έγγραφο εργασίας που λάβατε σήμερα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους προσκεκλισμένους μας και τους ε, εμπειρογνώμονες του πάνελ να λάβουν το λόγο. Απλώς δύο σχόλια πολύ σύντομα. Χρειάζεται και πρέπει να διασφαλίσουμε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού και ίσους κανόνες σε όλους τους τομείς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται προφανώς η δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Πρέπει να αποφύγουμε ε, μη ρεαλιστικές ε, προσεγγίσεις και τεχνητούς διαχωρισμό των διαφορών τομέων. Γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε ένα ενιαίο νομικό μέσο, το οποίο να καλύπτει όλου του τομεί και τι διαστάσει τη προστασία δεδομένων. Θέλω να είμαι ρεαλιστή και πραγματιστή στην προσέγγιση μου. Ε, μπορώ να κατανοήσω την ε, πορεία που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προηγουμένω την ε, περιέγραψε η Επίτροπο Ρέντινγκ. Όμω, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο επιμένουμε σε αυτό που θέλουμε να ονομάζουμε προσέγγιση δέσμη. Δηλαδή, ο κανονισμός και η οδηγία αντιμετωπίζονται σε μια κοινή δέσμη μέτρων ε, και ως προς την ουσία τους και ως προς τις πρακτικές τους ε, συνέπειες. Και το πώς βέβαια εμείς θα τις μελετήσουμε. Από αυτό το βήμα λοιπόν θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τα κρατη έκκληση να προχωρήσουν αμέσως ε, στην μελέτη της οδηγία. Ακούγονται φήμε, φτάνουν εδώ ειδήσει, έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει σκεπτικισμό, υπάρχει απροθυμία από κάποιου από τους ε, εταίρου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούν με την οδηγία. Επαναλαμβάνω, το Ευρωκοινοβούλιο ε, απευθύνει έκκληση να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση δέσμη, πακέτου. Και ε, εφόσον χρειαστεί θα υπερασπιστούμε ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Χωρίς λοιπόν άλλες καθυστερήσεις να δώσω το λόγο στον πρώτο μας ε, ομιλητή, τον Λόρδο Χένεϊ, με τον οποίο είχα την να μοιράζομαι μια μακρόχρονη φιλική σχέση. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές όταν ε, εργαστήκαμε σκληρά βέβαια για το κυπριακό ζήτημα και για την προσχώρηση της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ Δημήτρη, ε, συντονιστή. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας που ήταν ε, επανειλημμένες, πραγματικά είχαμε πολύ θετική συνεργασία. Δεν φαντάστηκα ποτέ να βρεθούμε όμως και σε ένα βήμα που θα συζητούμε το θέμα της προστασίας δεδομένων, ακόμη πιο περίπλοκο από αυτά που είδαμε στο παρελθόν. Χαίρομαι που έρχομαι στην ε, συνάντηση αυτή ω προσκεκλημένο και όχι ω εμπειρογνώμων απλώ. Ε, ε, αλλά έχω εργαστεί στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στην Υποεπιτροπή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ε, και η δική μα Επιτροπή μελέτησε και τον κανονισμό και την οδηγία πριν τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Θα συνεχίσουμε μάλιστα καθώ προχωρούν οι διαπραγματεύσει. Σε γενικέ λοιπόν γραμμέ, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει πλήρω μέρο στι διαπραγματεύσει αυτέ στηρίξαμε την απόφασή της. Και τα δύο αυτά νομοθετήματα εγείρουν ε, μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ αυτού που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ε, σε γενικές γραμμές όπως λέγονται τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των ενδιαφερομένων. Ε, υπάρχουν διαρκείς ενημερώσεις και διαρκείς επαφές με τον ιδιωτικό τομέα. Ε, ήδη πριν έρθω σε αυτή τη συνάντηση δέχτηκα πολλές ε, Είχα πολλές επαφές μαζί τους. Εδώ λοιπόν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το κάθε νομοθέτημα προχωρούν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον πρέπει να προσαρμόζονται βεβαίω τα κείμενα, ανάλογα με τι ανάγκε που ανακύπτουν και για να γίνουν πιο αποτελεσματικά ω προ την περιγραφή των στόχων. Τώρα, για την οδηγία, και επειδή αυτό είναι το βασικό ζήτημα της, αυτού του γύρου συζήτηση, για την συμπερίληψη των μέτρων προστασία δεδομένων στα γενικότερα μέτρα του ευρωπαϊκού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσε καλύτερο να προτείνει δύο ξεχωριστά νομοθετήματα. Αυτό μας φαίνεται ότι είναι μεν πραγματιστική αλλά και έγκυρη προσέγγιση. Η οδηγία θα επιτρέψει ένα επαρκές επίπεδο ευελιξία, ένα περιθώριο ελιγμού. Το κάθε κάτω μέλο θα μπορεί να λάβει υπόψη τι δικέ του ανάγκε. Όπω στη δική μα περίπτωση, λόγω χάρη, με το ξεχωριστό σύστημα του δικαίου μα, του Common ε, όταν θα πρέπει να μεταφέρουμε την οδηγία. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι η απόφαση πλαίσιο βέβαια που ήδη ισχύει είναι επαρκής αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην ε, πρόοδο της οδηγίας. Εγώ πιστεύω ότι η προτινόμενη οδηγία αποτελεί βελτίωση. Αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση πλαίσιο και ως προς πολλές πτυχές. Εάν τελικά εγκριθεί η οδηγία αυτή θα επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ότι οι διατάξεις της απόφασης πλαισίου Αυτή την απόφαση πλαίσιο, την εξέταση επιτροπή μου και στο παρελθόν είχε εκφράσει αμφιβολίε για, ε, για το κατά πόσο αποτελεσματική. Ε, οι διατάξει της οδηγίας δεν θα πρέπει να είναι πιο αδύναμες από ό,τι του κανονισμού και οι ελεγκτές ε, προσωπικών δεδομένων, μάλιστα ο ίδιος ο Βρετανός Επίτροπος για την Προστασία των Δεδομένων, επεσήμαναν το σημείο αυτό. Για επιχειρησιακούς βέβαια λόγους και επειδή το έργο των ε, διοκτικών αρχών κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα πρέπει η απόφαση αυτή και η δυνατότητα λήψης της απόφασης να ε, διασφαλιστεί. Επίσης κάποιοι ενδιαφερόμενοι και συνομιλητές μας εντόπισαν ασυνέπειε μεταξύ κανονισμού και οδηγία, ε, κυρίω ω προ τα εχέγγυα για την προστασία των δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα από τη μια και στον τομέα της επιβολής του νόμου από την άλλη. Πολλά από τα δεδομένα που συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς, όπως ε, για τις στατιστικές αναγνώρισης των επιβατόλογου χάρη, αυτά μπορεί να μεταφέρονται σε φορείς επιβολής του νόμου και κάποια οικονομικά στοιχεία πάλι για διοπτικού σκοπούς μπορεί να ε, μεταφερθούν για σκοπούς ε, καταπολέμησης της λεύκανσης προσόδων λόγου χάρη. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν πιο προσεκτικά και να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα στην περιγραφή τους. Τώρα, η ισχύουσα απόφαση πλαίσιο σε σχέση με την προτινόμενη οδηγία δείχνει ότι η πρώτη δεν καλύπτει την εσωτερική μεταφορά δεδομένων, ενώ η δεύτερη την καλύπτει. Κατανοώ ότι το αρχικό μέτρο το συμφωνησαν ομοφόνο ομοφόνος πολλά κράτη-μέλη, ε, αλλά έπειτα προτάθηκε η συμπερίληψη της εσωτερικής μεταφοράς. Η αρχική αυτή θυσία λοιπόν θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου να περάσει από απόφαση πλαίσιο το 2008. Εδώ όμως είμαι πιο αισιοδόξο από την Επίτροπο Ρέντινγκ. Για πρακτικούς και μονολόγους, ούτε καν ιδεολογικούς, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών εσωτερικής δηλαδή μεταφοράς ε, και διακριτικής. Η Επιτροπή μου δεν συμμερίζεται την άποψη που πολλέ φορέ εκφράστηκε από την κυβέρνησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θεωρούμε ότι δεν είναι πραγματιστικό ρεαλιστικό να κάνουμε τέτοια διάκριση μεταφοράς δεδομένων. εντός και μεταξύ των κρατών μελών δηλαδή. Η δική μας θεώρηση διαφέρει ελαφρώς. Επίσης, ένα ακόμη σχόλιο για πολλά από τα ευρωπαϊκά μέσα που αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων και την προστασία των δεδομένων, μεταξύ των οποίων η Europol, ο σχετικός κανόνας και η απόφαση Προύμ, όλα αυτά περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων τον ε, κανονισμό ε, θα υπερισχύουν οι τάξεις του κανονισμού σε σχέση με αυτές τις οδηγίες. Αυτό ε, βραχυπρόθεσμα φαίνεται λογικό, διότι η κάθε διάταξη έχει, θα έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις διάφορες επιχειρησιακές ανάγκες. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την νομική βάση και τη συνθήκη της Λισαβόνα. διότι τώρα έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να εξορθολογήσουμε την το κατακαιρματισμένο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Αυτό για την ώρα δεν φαίνεται να έχει επιχειρηθεί σε αυτή την ε, πρόταση οδηγίας. Οι διαπραγματεύσει βέβαια δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν προκειμένου να καλύψουν και αυτή την ανάγκη. Όμω η οδηγία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία διάταξη που να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών μετά τη θέση σε ισχύ διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ε, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσαν ε, να ε, εξεταστούν ανάλογα με το πώς έχει προχωρήσει και η οδηγία, πώς έχει υλοποιηθεί. Νομίζω ότι όλοι επιδιώκουμε ένα κοινό στόχο, ένα μια ψηφιακή ενιαία αγορά και για, αυτούς τους... για αυτές τις ανάγκες μπορούμε να επιδιώξουμε αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε πολύ τον Λόρδο Χάνι. Στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής φιλίας άλλαξε η Προεδρία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συμμετοχή σας και περνάμε στην Νταϊάννα Αλόνσο Μπλάς που είναι επικεφαλής ε, της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων στη Eurojust. Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων. Η κυρία Αλόνσο Μπλάς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ φοβούμαι ότι τα γερμανικά μου είναι πολύ ανεπαρκή και δεν μπορώ να σας απαντήσω στα γερμανικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ενώπιον σας και έχω την ευκαιρία να απευθύνω το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι διαδραματίζεται πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω πραγματικά να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και εσείς και εμείς. Πολύ συχνά μας θεωρούν ως εμάς, ως τους ανθρώπους που επιβάλλουν το νόμο. Εγώ δουλεύω στον τομέα της προστασίας δεδομένων από το 1994. Έχω συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές, τις Ολλανδικές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήμουν μέλος και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για πολλά χρόνια. Α, όλα αυτά πριν προσχωρήσω στη Eurojust. Και εν τω μεταξύ έχω πράγματι συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς τις ιδιαιτερότητες της ε, διεθνούς συνεργασίας σε ποινικά θέματα για να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα. Και η Eurojust και το κοινό ε, εποπτικό σώμα της Eurojust ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για το θέμα της προστασίας των δεδομένων και της πρόσβασης των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ατόμων, αλλά και για να πετύχουμε τους στοχούς μας. Δηλαδή, η επεξεργασία των δεδομένων είναι αδύρυτη ανάγκη για να πετύχουμε τους στόχους μας ως Eurojust. Και χαιρόμαστε ως Eurojust, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο που προτείνει έχει λάβει υπόψη της την ανάγκη να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες βάσει του τρίτου πυλώνα. Αυτοί οι ειδικοί κανόνες ε, δεν υφίσταται και δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο λόγω του διαφορετικού νομικού υπόβαθρου, αλλά και λόγω των διαφορετικών αναγκών ε, στην, ε, ε, στο πεδίο αυτό, λόγω των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων που υφίστανται. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν προβλέπει την αυτομάτως την ανάγκη να έχουμε ένα μέσο προστασίας δεδομένων. Στη συνθήκη της Λισαβόνας χρησιμοποιείται ο πληθυντικός αριθμός, ή αρχές και οι κανόνες. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ως προς το ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοχή, συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων εργαλείων, των διαφόρων μέσων, να έχουμε ένα ίδιο επίπεδο προστασίας. Μιλούμε για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και τον περιορισμό των καταχρήσεων. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια συνεκτική, συνολική προσέγγιση. Ω προ το σχέδιο οδηγίας, θεωρούμε ω Eurojust ότι είναι βελτίωση αυτό. Βελτιώνει το εφιστάμενο πλαίσιο, το έχει πει και η αξιότιμη επίτροπος κυρία ε, Ρέντιν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Ε, το ε, υφιστάμενο πλαίσιο ήταν πολύ περιορισμένο και γι' αυτό χρειάζεται αυτό το σχέδιο οδηγίας. Ωστόσο είναι γενικό λόγο το προτινόμενο τώρα η Eurojust συμμορφούνται με όλες τις γενικές αρχές ούτως ή άλλως που προτείνονται στο σχέδιο οδηγίας. Ωστόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δραστηριότητας της Eurojust, το σύστημα βάση του οποίου λειτουργεί είναι πολύ πιο λεπτομερές και προσφέρει ασφάλεια δικαίου. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οι δικοί μας κανόνες έχουν ειδικέ ασφαλιστικές δικλείδες για ειδικέ και ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα θύματα ή οι μάρτυρες. Έχουμε πολύ συγκεκριμένε προποθέσει. Πότε μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, για πόσο χρόνο μπορούμε να τα κρατούμε. Έχουμε κανόνε για την πρόσβαση στην πληροφορία. Έχουμε σαφ σαφέστατα όρια στην προστασία των δεδομένων. Μιλούμε για τη συμμόρφωση, για την υποχρέωση τα δεδομένα να είναι ενημερωμένα σχετικά και να μην είναι υπερβολικά σε ποσότητα ή σε περιεχόμενο. Όλα αυτά έχουν εφαρμοστεί, όλοι αυτοί οι κανόνες. Στο δικό μας σύστημα, το οποίο είναι και το μόνο σύστημα που χρησιμοποιούμε για να επεξεργαστούμε πληροφορίες. Συμπερασματικά λοιπόν πιστεύω ότι οι κανόνες μας ε, προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο οδηγίας. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι για λόγους ε, ευκρίνειας ορισμένοι πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερο όλα να καλύπτονται από το ίδιο σετ κανόνων. Αλλά και να το κάναμε αυτό δεν θα βελτιώναμε την προστασία των υποκειμένων. Αντιθέτως, η κατάστασή τους θα γινόταν πολύ πιο ασαφής, διότι θα βάζαμε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού να υπόκεινται σε πολύ γενικότερους κανόνες από αυτούς που θα τους χρειάζονται. Οι πιο συγκεκριμένοι κανόνες, οι πιο ειδικοί προσφέρουν περισσότερη προστασία στα άτομα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα δικαιώματα των, των ατόμων, κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία για τους ε, Ευρωπαίους βουλευτέ. Πολύ λεπτό το ζήτημα αυτό και πάντοτε η Eurojust εμπλέκεται στην αρχική φάση μιας ερευνητικής διαδικασίας όπου δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθούν δεδομένα χωρίς να τεθεί ε, σε κίνδυνο η έρευνα. Εμείς λειτουργούμε αναπερίπτωση, αναϋπόθεση ε, όπου δει και όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε παρέχουμε ή διαθέτουμε τις πληροφορίες αυτές. Όπου ε, είναι αυτό επικίνδυνο δεν το κάνουμε. Πολύ συχνά το δικαστήριο έχει επενέσει τον τρόπο με τον οποίο η Eurojust έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα και έχει προσεγγίσει τα θέματα αυτά και θεώρησε ότι όχι μόνο έκανε το καθήκον της ε, η Eurojust αλλά υπερεύει και αυτόν. Δηλαδή πήγαμε πολύ πιο πέρα από ό,τι ε, υποχρεωνο... Ε, μας υποχρέωναν οι κανόνες. Τα άτομα, τα δεδομένα των οποίων τα επεξεργαζόμαστε εμείς, σε καμία περίπτωση δεν στερούνται των δικαιωμάτων τους. Επομένως, η Eurobust έχει ένα στεναρό σύστημα προστασίας δεδομένων το οποίο έχει προσαρμόσει στην εντολή που έχει λάβει και ε, το σύστημα αυτό το επιβλέπει το κοινό εποπτικό σώμα και οι ε, υπεύθυνοι ε, που είναι στις διευθυντικές θέσεις. Εμείς συνεργαζόμαστε σε ε, δικαστικές διώξεις, έρευνες, αστυνομικές έρευνες, πράγματα που διενεργούνται σε και σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων έχουν την αρμοδιότητα, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων δεν είναι αρμόδιες για να ε, ε, αποφανθούν περί της επεξεργασίας των δεδομένων από το δικαστήριο το κοινό εποπτικό στόμα τα παρακολουθεί όλα αυτά και σέβεται την, ε, τον ειδικό χαρακτήρα της δικαστικής εξουσίας. Θα ήθελα τώρα εν συντομία να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Γιατί λειτουργεί τόσο καλά το δικό μας κοινό εποπτικό σύστημα. Πρώτον έχουμε την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Το κοινό εποπτικό σώμα ε, απαρτίζεται και από εκπροσώπους εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και από δικαστές. Είναι όλοι ανεξάρτητοι λειτουργούν εν πλήρη ανεξαρτησία λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δουλειάς τους. Δεύτερον, είναι πολύ αποτελεσματικό. Τρία ερετά μέλη ε, συνεδριάζουν τέσσερις ή πέντε φορές το χρόνο στα γραφεία της Eurojust. Στοιχίζει και όλα έχουν τιμή σήμερα ε, και πρέπει να αναφερθεί τιμή σε καιρούς ε, κρίσης, στοιχίζει λιγότερο από 40.000 ευρώ το χρόνο και πάντοτε καλούμε τα κράτη-μέλη να ε, εμπλακούν στην διαδικασία. Είναι μια γρήγορη και καθόλου δίσκαμπτη διαδικασία. Ε, κάνει επίσης το Κοινό Εποπτικό Σώμα ελέγχους και επιθεωρήσεις επιτόπου, μαζί με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Έχουμε κοινέ επιχειρήσεις. Συν τις άλλες, έχουμε πλήρη διαφάνεια. Ε, το Κοινό Εποπτικό Σώμα έχει στο σελίδα, βλέπετε εκεί και βρίσκεται όλες τις ενημερώσεις, το, ο, τις εκθέσεις και το καθεξής. Και τέλος, και πολύ σημαντικό, οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές για τη Eurojust. Το κοινό ευρωπτικό σώμα λοιπόν ε, έχει αυτή τη δυνατότητα. Και κάτι το οποίο είναι σημαντικό νομίζω για τα εθνικά κοινοβούλια είναι το εξή. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε εμείς από τη Eurojust μας έρχονται από τα κράτη-μέλη και επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Επομένως οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι λογικό να εμπλέκονται στην εποπτεία και την υποθεώρηση αυτό αυτών. Και εξού και ε, έχουμε εκπροσώπους των κρατών μελών ως μέλη. Ως Eurojust δεν είμαστε κατά της ενισχυμένης συνεργασίας. Θέλουμε μόνο να δηλώσουμε ότι έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί καλά, που είναι αποτελεσματικό, που ταιριάζει στις ανάγκες μας ως υπηρεσία και που συμμορφούνται με τους κανόνες για την υψηλή ε, προστασία ε, των ατόμων και για την αυξημένη ασφάλεια δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Ας μην επισκευάσουμε κάτι το οποίο δεν έχει χαλάσει και δεν χρειάζεται επιδιόρθωση, ούτε επισκευή. Ας διασφαλίσουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ε, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν θα μακρηγορήσω. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι έχουμε φέρει πολύ υλικό εδώ για τη δουλειά της Eurojust στον τομέα Τη προστασία δεδομένων έχουν μοιραστεί τα φυλάδια, δεν έχουμε άλλα αντίτυπα, αλλά αν θέλει κάποιο μπορεί να μου το πει να του το στείλω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και ευχαριστώ και την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη στήριξη που μα προσφέρετε στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ε, συνεισφορά σας. Και τώρα από τον ένα ευρωπαϊκό οργανισμό σε έναν άλλο. Μια ευρωπαϊκή υπηρεσία μάλλον στην άλλη. Ο κύριο Ντρούερ, υπεύθυνο Προστασία δεδομένων και ο κύριος Μάνιξ που μάλλον θα παρέμβει μετά. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ντρούερ από την Europol. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή μου να σας απευθύνομαι σήμερα ω υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων από την Europol και δίπλα μου είναι ο κύριο Όμαν από το Τμήμα Επιχειρήσεων τη Europol. Είναι στη διαθεσή σα εφόσον στη συνέχεια έχετε ερωτήσει για το επιχειρησιακό έργο τη Europol. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι από τι βασικέ δραστηριότητε τη Europol. Η είναι κύρια δραστηριότητα της Europol ώστε να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ε, προστατεύσουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρομοκρατικές επιθέσεις και το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει ένα πλήρες ε, σύνολο κανόνων που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της προστασίας των δεδομένων. Όλοι οι κανόνες αυτοί είναι συνάδουν με του γενικότερου κανόνε τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Απλώ στην αστυνομική συνεργασία ε, έχουμε να κάνουμε ευαίσθητο στο θέμα που απαιτεί ειδική προσοχή. Οι ιδιαιτερότητε του τομέα αυτού δεν έχουν να κάνουν μόνο με την διάρθρωση τρίτου πυλώνα που είχαμε λόγω των προηγουμένων ευρωπαϊκών συνθήκων αλλά προκύπτουν και από τη δήλωση 21 της συνθήκης ε, της Λισαβόνας. τα ευάλωτα δεδομένα, εφόσον ύποπτοι μπορεί, θύματα ή μάρτυρες μπορεί να εμπλέκονται σε ερευνητικές δραστηριότητες, ε, χρήζουν ιδιαίτερη προστασίας. Αυτά συνήθως τα διαχειρίζεται ακριβώς η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, η Europol. Τα συστήματα ε, ενημέρωσης επίσης που χρησιμοποιούμε και πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικά όπως το, η αρχή του σχεδιασμού που έχουν ακολουθήσει και η Eurojust, όπως ανέφερε η κυρία Αλόνσο και η Europol. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη τις ειδικές ανάγκες των χωρών και τα δικαιώματα των πολιτών σε συγκεκριμένες χώρες σε διεξαγόμενες έρευνες. Υπάρχουν τώρα αυστηρές προδιαγραφέ για το πότε μπορούν να τύχουν επεξεργασίε στα δεδομένα και για χρονικέ προθεσμίε. Για την κράτηση επίση των δεδομένων και συστηματική αναθεώρηση τη συμβατότητα των προσωπικών δεδομένων με, υπόλοι... με του υπόλοιπου κανόνε. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, εύστοχα και όχι υπερβολικά. Όλοι οι, κανόνες όλοι οι κανόνες αυτοί διέπουν τις δραστηριότητες ε, προστασίας των δεδομένων της Europol. Αυτό προκύπτει και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για οποιοδήποτε νέο σύστημα θεσπίσουμε βάση της, του άρθρου 10 της απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση της Europol. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πολύ συχνά απευθύνονται στην Europol και θέλουν να ξέρουν ποια στοιχεία τους αφορούν ε, στην επεξεργασία που κάνουμε στο σύστημά μας. Πολλά αιτήματα που λαμβάνουμε από τους πολίτες, ε, όπως το 2006, ε, ήταν ολιγάριθμα. Το 2006 μάλλον είχαμε 19 μόνο τέτοια αιτήματα, φέτος έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 600. Η εξέταση τέτοιων αιτημάτων και στην ίσια με τα κράτη-μέλη είναι επίσης βασική μέρημνα της Europol πρόσθετη εγγύηση είναι ότι μπορεί από το κοινό ε, εποπτικό όργανο να ζητήσει βοήθεια ο κάθε πολίτης και να ζητήσει την επεξεργασία δεδομένων ε, από την Europol πάντοτε σύμφωνα και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ίδρυση της υπηρεσίας. Τώρα, εξορισμού, ο Ευρωπαίος πολίτης λαμβάνει απάντηση από την Europol ευθύς αμέσως στο αίτημά του μαθαίνει τι αφορούν τα δεδομένα, εάν υπήρξε συλλογή και αν ήταν αυτή αναγκαία. Τώρα ένα άλλο ζήτημα είναι εγγυήσει που ισχύουν στη συνεργασία μας με τρίτα μέρη. Η Europol μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με τρίτα μέρη μόνο βάσει επιχειρησιακής συμφωνίας. Υπάρχει ένα παρόμοιο σύστημα εδώ όπως και στην Eurojust. Δηλαδή πρέπει να παράσχουμε στο Συμβούλιο έκθεση αποτίμησης προσωπικών δεδομένων. Εκεί βλέπουμε δηλαδή τι νομοθεσία επικρατεί στην τρίτη χώρα και τι διοικητικές πρακτικές ισχύουν στις αστυνομικές και δικαστικές τους αρχές προκειμένου να γίνει μελλοντικά και εταίρος μας, συνεργάτης μας. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε μια διεξοδική, όπως έλεγα, μελέτη που επιτρέπει στους εμπλεκόμενους φορείς να αποτιμήσουν την κατάσταση προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ε, λόγω τρίτη χώρα. Οι διατάξεις μας για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι επίσης αρκετά λεπτομερείς και αφορούν όλες τις διεκτικές αρχές αυτής της τρίτης χώρας. Τώρα, για το άρθρο 16 της συνθήκης της Λισαβόνας και τη σχετική συνεργασία, κάθε δραστηριότητα χρήσης δεδομένων θα πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό συμβαίνει και στη Europol με συγκεκριμένο σύστημα επιθεώρησης από το 1999. Η υλοποίηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων σε μια πρώτη φάση την χάνει επιθεώρηση από τον υπεύθυνο προστασία δεδομένων εντό Europol και μετά από την κοινή υποπτική αρχή. Εκεί ε, συμμετέχουν ε, υπάλληλοι από τι 27 εθνικέ αρμόδιε αρχέ και ε, οι αρμόδιοι που ασχολούνται με τα θέματα της Europol. Οι, εκ, οι αναλυτικές εκθέσεις που αποστέλλονται από το Europol προς τα κράτη-μέλη προκύπτουν ακριβώς από την μελέτη των επιχειρησιακών μα δραστηριοτήτων, της συλλογή δεδομένων και της δραστηριότητας ε, μελέτης τους. Από τη στιγμή που τα δεδομένα ε, συλλέγονται από τα κράτη-μέλη, αποστέλλονται στη Europol για να μπορέσει να φέρει πέρα στα καθήκοντά τη, αναλύονται από τη Europol, τελικά φαίνεται ότι από την πορεία αυτή καταλήγουν στα κράτη-μέλη, ώστε οι εθνικέ αρχέ παρακολούθηση να τα εξετάσουν και να μπορέσουν να έχουν συνομιλία και επικοινωνία με την αρχή που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της Europol. Ε, το σύστημα λοιπόν της Europol ε, λειτουργεί αποτελεσματικά. Είναι αποτελεσματικός ο μηχανισμός που σήμερα εφαρμόζεται. Προστατεύονται οι πολίτες, τα άτομα για τα οποία συλλέγονται δεδομένα, ακόμη και να εμπλέκονται σε διεξαγόμενες αστυνομικές έρευνες. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα σε αυτή τη φάση θα πρέπει προσεκτικά, να, να σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπερθούν βελτιώσει στη διαχείριση των δεδομένων που αφορούν του πολίτε από την Europol στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζουέ. Και τώρα από την πρακτική στην επιστήμη. Από το Ινστιτούτο Max Planck για το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο στο Φράιμπουργκ, η κυρία Έλς Ντεμπούσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που με κάλεσε σήμερα σε αυτή την ε, ε, διάσκεψη. Ε, νομίζω ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία σήμερα να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε μια συγκεκριμένη πρόκληση στην επιβολή του νόμου που για μένα είναι πολύ σημαντικό που είναι η αρχή της προστασίας του, του περιορισμού του σκοπού. Ο στόχος συλλογής δεδομένων είναι για την συλλογή πρόληψη, διερεύνηση, ανείχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων και υπάρχουν και δεδομένα τα οποία συγκεντρώνουν ιδιωτικές εταιρείες. Καταγράφονται συμπεριφορές των πολιτών όπως και αγοραστικές συμπεριφορές με σκοπό την ανείχνευση του αν ένα συγκεκριμένο άτομο προγραμματίζει κάποιο ποινικό αδίκημα. Αυτό το οποίο είναι κέρια σημασίας πιστεύω είναι η διάκριση μεταξύ τριών σκοπών, τριών τύπων σκοπού. Καταρχήν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο μιας ποινική διερεύνησης. Στη δεύτερη ομάδα υπάρχουν δύο είδη σκοπών που είναι διαφορετικοί, δηλαδή προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται για άλλους σκοπούς, αλλά είναι αντικείμενο επεξεργασίας για την διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων και μπορεί να είναι συμβατός ή μη συμβατός αυτός ο σκοπός. Για τον αρχικό σκοπό που αναφέραμε, Βλέπουμε ότι στο άρθρο 4 ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι επαρκή σχετικά και όχι υπερβολικά. Εδώ θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε νομίζω με πιο έντονο τρόπο. Γιατί η ελαχιστοποίηση των δεδομένων είναι μια αρχή που θα έπρεπε εδώ να εμφανιστεί πολύ πιο στεναρά αυτό το τμήμα της πρότασης ε, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα ε, να εκφράζεται σαφέστερα η αναγκαιότητα. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται για το σκοπό ποινική δίωξης ε, ίσως πρέπει να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται της πρόληψης διερεύνησης ανείχνευσης ή δίωξης για, μια, για ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα ή για ένα συγκεκριμένο άτομο. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα είναι σύμφωνο αυτό και με τη σύσταση 97 του Συμβουλίου της Ευρώπης που το βλέπουμε να προκύπτει σε αρκετά σημεία της πρότασης. Τώρα, για την άλλη ομάδα ε, σκοπών, μπορούμε να δούμε αν είναι συμβατή με το στόχο μας ή όχι. Ένα ε, ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε ορισμός για το τι αποτελεί συμβατό σκοπό. Εδώ νομίζω βρισκόμαστε σε μια στιγμή που πρέπει να υποφεληθούμε τις ευκαιρίες για να το συζητήσουμε και εποφελούμε σήμερα να κάνω μια προσπάθεια να ορίσουμε τι είναι συμβατός σκοπός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό, το ξέρω, αλλά κάποιες ενδείξεις για το τι είναι συμβατός σκοπός θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην πρόταση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προτείνω έναν ορισμό και θα πρέπει να συμπεριληφθεί το γεγονός ότι ένας συμβατός σκοπός πρέπει να έχει κάποια λειτουργικά ισοδύναμα Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποια σύγκληση, να μην είναι απλό σχετικό σκοπός, αλλά κάτι περισσότερο. Ε, Μία δεύτερη προϋπόθεση για να είναι συμβατό ο σκοπός είναι ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον προβλέψιμο από την πλευρά του υποκείμενου στη συλλογή δεδομένων. Και θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για συμβατούς σκοπούς εάν, και πάλι εδώ υπάρχει προϋπόθεση της αναγκαιότητας, εάν είναι αναγκαία για ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα ή για την έρευνα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο. Όταν λοιπόν ορίσουμε τι είναι συμβατός σκοπός, θα είναι πιο εύκολο να ορίσουμε τι είναι ασύμβατος σκοπός. Και εδώ συμφωνώ απολύτω με την άποψη που δημοσιεύθηκε από τον, Ευρωπαίο, από τον επόπτη ε, δεδομένο. Στο άρθρο 7 της οδηγίας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει χωριστή παρέκκληση από την αρχή του περιορισμού του σκοπού. Το άρθρο 7 λέει ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να παρεκκλίνουμε. Δηλαδή θεωρεί ένα καθήκον που βασίζεται με τους σκοπούς του άρθρου 1 της οδηγίας όπως αναφέρονται εκεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής παρέκκληση από την αρχή του περιορισμού του σκοπού. Πρέπει να είναι κάτι το νόμιμο και θα, νομότυπο και θα πρέπει να είναι και απαραίτητο, αναγκαίο για την έρευνα ενός συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος ή συγκεκριμένου ατόμου. Και μια τελευταία παρατήρηση για κάποιες άλλες διακρίσεις, τις οποίες θεωρώ θετικές. Χάρηκα πολύ που τις βλέπω μέσα στην πρόταση αυτή. Καταρχήν η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών βαθμών ακριβίας και αξιοπιστίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν μιλάμε για ποινικέ έρευνες, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ στοιχείων ή εκτιμήσεων και πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιστήρια σε μια ποινική δίκη. Και εδώ πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθούμε στα δικαιώματα, στο δικαίωμα δίκαιης δίκης και πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βαθμών ακρίβειας και αξιοπιστίας. Η Europol μπορεί να είναι χρήσιμη σε αυτό γιατί έχει πίνακα του τι είναι επιβεβαιωμένα και μη επιβεβαιωμένα στοιχεία. Δεύτερον, διάκριση κατηγοριών υποκείμενων ε, στην συλλογή δεδομένων και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση και χαίρομαι που υπάρχει μια τέτοια διάκριση και θα ήθελα και εδώ να αναφέρεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη γιατί εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε κυρίως για υπόπτους, αλλά εκτός από τους υπόπτους υπάρχει και μια μεγάλη κατηγορία ε, των μαρτύρων και υπάρχει και μια μεγάλη κατηγορία παιδιών, επομένως θα πρέπει να προστατεύονται. Η Eurojust έχει ε, συμπεριλάβει αυτές τις κατηγορίες με πολύ καλή διάκριση ε, στους κανόνες της για την προστασία των δεδομένων. Αυτά λοιπόν για την αρχή της, του περιορισμού του σκοπού. Και θα ήθελα να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έκανε κατά τη σύνταξη της πρότασης αυτής. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να ρυθμιστούν περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντεμπουσέ. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Άννα Φίλντερ από την Privacy International στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω ε, αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Πράγματι, οι περισσότερες συζητήσεις των εμπλεκόμενων μερών στρέφονται γύρω από τον κανονισμό και λιγότερο γύρω από την οδηγία, ενώ στην πραγματικότητα οι πολίτες ενδιαφέρονται κυρίως για το σύνδρομο του μεγάλου αδερφού και για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτά από τις δημόσιες διοκτικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής πολιτικών ελευθεριών για την πρόσκληση που μας απίφθεναν. Η Privacy International ε, λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια. Είναι ένας ιδιωτικός φιλανθρωπικός οργανισμός και στόχο έχει να υπερασπιστεί την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας παντού στον κόσμο ε, έναντι της εισβολής ε, στην ιδιωτική σφαίρα και στην ιδιωτικότητα των κυβερνήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Βεβαίως, τα τελευταία τρία χρόνια στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα αναθεώρησης ε, του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου ώστε να έχουμε μια συνεκτική και υψηλού επίπεδου προστασία προσωπικών δεδομένων. Στην παρουσίασή μου θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις ή και για τα εγχώρια ζητήματα και κατά δεύτερο λόγο θα αναφερθώ στο περιεχόμενο της οδηγίας και πώς ε, συντεριάζεται με το περιεχόμενο του κανονισμού ε, παρουσιάζοντας το πρίσμα, την οπτική γωνία των πολιτών και της κοινή γνώμης. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πλαίσιο προστασίας δεδομένων πρέπει να ισχύει και για τις διασυνοριακές διαβεβάσεις και για την εγχώρια επεξεργασία σε έναν ε, ιδανικό κόσμο και συμφωνώ και με τον κύριο Δρούτσα υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε επιτάπητος να είχαμε μόνο μία πρόταση για την προστασία δεδομένων, μία, μόνο, μία και μόνη νομική πρόταση ε, για όλα με τους κατάλληλους κανόνες και τους κατάλληλους περιορισμούς ανακλάδο και Η πλειονότητα των κρατών μελών έχουν ε, εφαρμόσει ε, την οδηγία για την προστασία των δεδομένων παντού πολύ συχνά προβλέποντας εξαιρέσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου. Ακόμα και σε χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία και οι κάτω χώρες, όπου οι αρχές επιβολής του νόμου υπάγονται σε άλλη νομοθεσία, η ίδια συνταγματική αρχή συνεχίζει να ισχύει. Αυτή που ε, βρίσκεται πίσω από το, τους νόμους για την προστασία δεδομένων. Τώρα όμως έχουμε μια ξεχωριστή οδηγία η οποία ε, θα ισχύει από μόνη της. Αυτό προτείνεται και έτσι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν δύο νομοθετήματα στη τιμή του ενός. Αυτό θα επιφέρει πάρα πολύ μεγάλη περιπλοκότητα και δεν θα γίνει εφικτό να πετύχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων για τους πολίτες ανα πάσα στιγμή και σε κάθε συνθήκη. Αναπόφευκτα, η ενσωμάτωση της οδηγίας στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες θα οδηγήσει στον κατακαιρματισμό τον οποίο ακριβώς θέλει να αποφύγει αυτό το υποτιθέμενο νέο νομικό πλαίσιο. Τελικά μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε μία και ενιαία γενική νομοθεσία για, τον την προστασία των δεδομένων και 27 τελικά διαφορετικά καθεστώτα που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς των αρχών επιβολής του νόμου. Και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών όταν οι πληροφορίες που τους αφορούν τις μοιράζονται μεταξύ τους διάφορες χώρες. Και ε, δεδομένα που συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς όταν χρησιμοποιούνται ε, από αρχές επιβολής του νόμου ε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όλο και συχνότερα και θα δημιουργήσει όλο και περισσότερα προβλήματα με την υφιστάμενη αυτή πρόταση. Επεξεργάζομαστε τα δεδομένα για γενικούς σκοπούς ή, ή το κάνουν οι ιδιοκτικές αρχές πώς δεν θα καταστρατηγηθούν τα δικαιώματα των ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταλήξει σε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία ε, αυτών για τους οποίους γίνεται έρευνα, τους υπόπτους και τους κατηγορημένους. Το 2009 ένας οδικός χάρτης υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και προτείνονται νομοθετικά μέτρα πάνω σε διάφορα θέματα. Ε, νομική συμβουλή, δικαίωμα στη μετάφραση, προστασία ε, ευπαθών ε, υπόπτων, υπόπτων σε δύσκολη κατάσταση και Σε αυτό το οδικό χάρτη δεν περιλαμβάνεται η προστασία των δεδομένων, θα έπρεπε όμω να είχε συμπεριληφθεί, ούτω ώστε να πετύχουμε το στόχο τη αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή μια δικαστική απόφαση που ε, υιοθετείται σε μια χώρα να ε, αναγνωρίζεται σε μια άλλη. Μεταξύ ε, άλλων αυτό είναι ο βασικός λόγος για την προτινόμενη οδηγία η οποία θα πρέπει να ισχύσει και στο εγχώριο επίπεδο η επιβολή του νόμου δεν έχει να κάνει μόνο με τους ε, εγκληματίες του ποινικού δικαίου, τους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους. Οι διοκτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν επίσης να κάνουν με θύματα, με μάρτυρες, με διαφόρους άλλους που έχουν εμπλακεί στα, δίκ, δίκτυα των ε, ερευνών. Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική και αυξάνει τον κίνδυνο να διακινδυνεύσουν διάφορα πράγματα διάφοροι πολίτες. Έχουμε ε, ελέγχους DNA και ελέγχους βιομετρικών δεδομένων οι οποίοι γίνονται πλέον ως ρουτίνα και έτσι άνθρωποι μπαίνουν σε πολύ δύσκολες και λεπτές ε, ε, συνθήκες και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 50 εκατομμύρια άνθρωποι π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ε, τα δεδομένα τους διατηρούνται και διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκ των οποίων ενδεχομένω 6 εκατομμύρια είναι παντελώς αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση ε, με τις υποθέσεις για τις οποίες γίνεται έρευνα. Το 20% είναι η γενικότερη εκτίμηση. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό οι διατάξει τη προτινόμενη οδηγία να είναι αρκετά στεναρέ, να είναι εναρμονισμένε με αυτέ τι διατάξει του προτινόμενου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Γιατί έτσι όπω έχουν διατάξει αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο ισχυρέ. Θεωρούμε ότι στην προτινόμενη οδηγία οι αρχέ για την επεξεργασία των δεδομένων είναι λιγότερο φιλόδοξε, είναι περισσότερο ε, περιορισμένες από αυτές στον κανονισμό τα δικαιώματα των ε, κατόχων των δεδομένων αυτών ε, τα προστατεύουμε πολύ λιγότερο από ό,τι στον κανονισμό. Οι ελεγκτές έχουν λιγότερες εξουσίες και αρμοδιότητες και λιγότερο ισχυρές εξουσίες για παράδειγμα, η αρχή του περιορισμού του σκοπού που ανέφερε εκτεταμένα ε, προηγούμενο συνάδελφο. Λέει ο κανονισμός ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο δυνατό. Ενώ στην οδηγία η διατύπωση είναι όχι υπερβολικά. Δεν λέει θα πρέπει να περιορίζεται, αλλά λέει όχι υπερβολικά. Έχει διαφορά ο ένα όρο από τον άλλον. Ε, στη συνέχεια, ε, η έλεγχη μπορεί να είναι λιγότερο διαφανής, ε, να είναι πιο βραδία η απάντηση, να μην υποχρεούνται τόσο πολύ προς απάντηση. Τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν νομοθεσία που ε, θα χαρακτηρίζει με το χύψη τρόπο ολόκληρες ομάδες προσωπικών δεδομένων, ολόκληρες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Δεν απαιτείται από τους ελεκτές να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με την προτινόμενη οδηγία και δεν γίνεται καμία αναφορά στα παιδιά στην οδηγία. Για σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, πολύ πιο αδύναμη η διατύπωση στην οδηγία. Σε, σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν, στηρίζουμε αυτή την πρόταση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων για να φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αλλά μένει με πολλή απόσταση να διανύσουμε για να τα καταφέρουμε αυτά. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι νομοθέτες, οι αιρετοί ε, πολιτικοί ε, από όλες τις γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα συμμορφούνται με τους ίδιους κανόνες για την προστασία των δεδομένων όπως και οι υπόλοιποι. Και κατά δεύτερο λόγο, οι κανόνες να ισχύσουν παντού, εγχώρια και ε, στο εξωτερικό, και τρίτον, όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε, να τα επεξεργαστούμε ως πακέτο, ως σύνολο, να τα εγκρίνουμε την ίδια στιγμή και να μην παραχώσουμε την οδηγία κάτω από το χαλάκι ε, και να τελικά να την ξεχάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ήσασταν η τελευταία ομιλητρία σε αυτό το πάνελ, οπότε πάλι έχουμε ένα γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. δεν είναι πάντοτε απλό ε, οι πολιτικοί ή οι νομοθέτες να ακολουθούν ε, την σωστή μέση οδό μεταξύ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και της προστασίας αυτών. Υπάρχει πάντοτε το θέμα του πόσο μπορεί να προχωρήσει το κράτος και ε, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Όλα αυτά τα θέματα είναι προς συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τώρα τις ερωτήσεις, ξεκινώντας από τον συνάδελφο Άλβαρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που περιγράψατε, ε, σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο, είναι ακριβώς το μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που μας ε, διαχωρίζει από χώρες που θα χαρακτηρίζονταν ως μπανανίες. Άκουσα τη συνάδελφα από το ε, Max Planck και από την Privacy International και άκουσα ε, και το γενικότερο πλαίσιο το οποίο περιγράφουν υπάρχει γενικότερη προβληματική του δημοσίου δικαίου. Ε, Τέθηκε το ερώτημα του τι είναι συμβατό, ποιοι σκοποί είναι συμβατοί. Ο κανονισμός παραπέμπει και στην οδηγία, γι' αυτό πρέπει να δούμε ποια είναι η σωστή ε, ε, νομική τάξη. Και η δημόσια ασφάλεια είναι μια έννοια την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η ερώτησή μου αφορά περισσότερο τις υποχρεώσεις που θέτει ο κανονισμός ε, προς τους ιδιώτες υπάρχουν ε, υποχρεώσεις επί των ε, δημοσίων αρχών και νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε σαν κριτήριο ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να υπάρχει νομιμοποίηση. Θα πρέπει να δούμε τις υποθέσεις ε, νομικών, εκπροσώπων του κλήρου κλπ. Θα δούμε και τι μπορεί να γίνει για τους δημοσιογράφους. Και ε, κατά πόσον η ακρίβεια των δεδομένων μπορεί να είναι εξασφαλισμένη και στο έγγραφο του εισηγητού υπάρχει ε, κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε ε, επιτύχει κάποια εργαλεία από το ΠΡΟΥΜ και πρέπει να δούμε πώς θα χειρίζονται τα διάφορα κράτη-μέλη και αν μπορούν αυτά να τα χρησιμοποιήσουν και άλλα κράτη-μέλη. Τα βασικά ερωτήματα λοιπόν προς το πάνελ είναι αν είναι βιώσιμο να πούμε, αν μπορεί κανείς να το πει, ότι δεν θα παρεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές αν δεν υπάρχει ε, δεν, δεν το ζητάει κάποιος ε, νομικός, αν δεν υπάρχει νομική επίκληση. Δεν θα υπάρχει ε, κάτι αντίστοιχο για τους ε, δικηγόρους και άλλες παρόμοιες ε, κατηγορίες. Και τι γίνεται με, τις, με τα διάφορα θεσμικά εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδερ. Και δίνω το λόγο τώρα. Ελπίζω να πω σωστά το όνομά σας. Κυρία Μπατήλ. Μπατέτ. Σας ευχαριστώ. Σχεδόν τέλεια το προφέρατε το όνομα μου. Μία παρατήρηση. Κάτι που ενδεχομένως δεν αφορά απλώς τη σημερινή συζήτηση και δεν είναι και καταλληλότερη διάσκεψη για να θέσω ένα τέτοιο ζήτημα. Όμως μετά την ομιλία της κυρίας Φίλντερ, η οποία εκπροσωπεί την Privacy International, Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σχέση έχετε με την Transparency International. Πρόκειται για δύο ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες, κατά τρόπο παρόμοιο. Γίνεται πολλή λόγος για την προτινόμενη οδηγία. Όταν ε, φτάνουν πολλές φήμες στα αυτιά των πολιτών, όταν πολλής λόγος γίνεται για τον ιδιωτικό βίο, αυτό συσχετίζεται απευθείας με ένα θέμα που σε κοινωνικό επίπεδο ίσως να μην είναι τόσο ε, δημοφιλές, αλλά πρόκειται για την ανάγκη διαφάνειας. Διαφάνεια στη λειτουργία των δημόσιων φορέων. Αυτά είναι δύο ζητήματα που πρέπει να οδεύουν παράλληλα. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρέπει να προσφέρονται οι ίδιες εγγύησεις, η προστασία του ιδιωτικού βίου και το δικαίωμα στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση κατά τρόπο παρόμοιο. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες. Και μάλιστα σε μία φάση όπως η τωρινή μια φάση όπου η αξιοπιστία μας είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να ακολουθούμε προσέγγιση διαφανέστερη, πιο ανοιχτή προς τους πολίτες. Μας, μας ζητάτε να βρούμε αποκρίσεις σε προβλήματα καυτά της επικαιρότητα, όπως η οικονομική κρίση. Γι' αυτό μας ζητάτε να λειτουργούμε και με τρόπο πιο ανοιχτό, πιο διαφανή. Γιατί εδώ ακριβώς ε, διακυβεύεται η αξιοπιστία μας. Για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πέραν αυτού του πακέτου, της δέσμης δηλαδή μέτρων του κανονισμού και της οδηγίας, για την προστασία του ιδιωτικού βίου, ίσως θα πρέπει να σκεφτούν ότι χρειάζεται και κάτι ακόμη για να συμπληρωθεί το πακέτο, η διαφάνεια του δημόσιου βίου ή της λειτουργίας των δημοσίων φορέων. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφο Μπρίγκετ Τσίπελ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αρχικά δεν ήθελα το λόγο, Νομίζω ότι θα υπήρχαν ε, πολλές συνεισφορές από εθνικά κοινοβούλια. Ε, θα ήθελα όμως να υποφεληθώ της ευκαιρίας ε, για να μιλήσω για ένα σημείο το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά αντιφατικό. Η κυρία Ρέντινγκ στην παρέμβασή της μίλησε για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης χρησιμοποιούμε πάντοτε μια διατύπωση στο πλαίσιο της συνεργασίας ότι βασίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι υπάρχει εμπιστοσύνη ή πρέπει να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ότι θα πρέπει οι πολίτε να έχουν εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και στο πώ θα χειριστούν οι επιχειρήσει ή το κράτο τα στοιχεία του, αλλά οι πολίτε θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και στο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Και το λέω έχοντας συνείδηση του τι λέω. Όταν πρόκειται για τα δικαιώματά τους, οι πολίτες δεν έχουν κατανόηση για το ότι τα δικαιώματά τους είναι αντικείμενο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα σε ορισμένα κράτη-μέλη καλύτερα και σε άλλα κράτη-μέλη χειρότερα. Οι πολίτες θέλουν να έχουν σωστή προστασία των δικαιωμάτων τους και γι' αυτό νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι καλό θα ήταν και στον τομέα της συνεργασίας, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας να έχουμε κανονισμό. Ακριβώς διότι χρειαζόμαστε εξίσου καλά και υψηλά πρότυπα σε όλα τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε τα δικαιώματα των πολιτών να είναι αντικείμενο επεξεργασίας με ίσο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως κατηγορούμενος, ως θύμα ή ως μάρτυρας, μπορεί να εμφανιστώ και σε άλλο κράτος μέλος και να εμπλακώ σε μια ποινική διαδικασία και θα ήθελα να είμαι εξασφαλισμένη ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα είναι αντικείμενο λογικής και ορθής επεξεργασίας. Και όταν τα δεδομένα κυκλοφορούν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο και θα πηγαίνουν μόνο στις αρχές που ασχολούνται με την δικαστική υπόθεση και θα μένουν εκεί και δεν θα καταλήγουν στα μέσα ενημέρωσης ή δεν θα καταλήγουν στους αντιδίκους ή σε κάποιον ε, όπου θα, ήταν, ε, ε, θα διακινδύνευα για τα προσωπικά μου συμφέροντα. Αυτό είναι λοιπόν μια προϋπόθεση που πρέπει να έχουμε στις ε, συζητήσεις μας. Και γι' αυτό θα πρέπει στο θέμα των ε, δεδομένων και της ανταλλαγής των δεδομένων ε, να το έχουμε υπόψη αυτό για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία γιατί πρόκειται για την προστασία των δεδομένων των πολιτών και θα πρέπει να διευκρινίζεται ποιο είναι ε, το δημόσιο συμφέρον. Η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να είναι εγγυημένη ακριβώς διότι θέλουμε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και μεταξύ των αρχών αλλά και μεταξύ των πολιτών και των αρχών. Υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν σε αυτό το τομέα και υπάρχουν και διαφορετικές νοοτροπίες στις διάφορες χώρες. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, αλλά τα δικαιώματα θα πρέπει παντού να είναι αντικείμενο σωστής προστασίας. Και νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να το επιτύχουμε για την προστασία των δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν δώσω το λόγο στους εκπροσώπους εδώ στο Προεδρείο, να δούμε αν υπάρχει και κάποια ερώτηση, αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Από τα Εθνικά Κοινοβούλια ίσως δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους ε, συμμετέχοντες στο Προεδρείο, ξεκινώντας από τον Λόρδο ε, Χένι. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και φαίνεται πόσο καταπληκτικό είναι το θέμα. Υπάρχουν διαφορετικές πιέσεις μεταξύ της προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων και της ε, αυξανόμενης ανάγκης ευρωπαϊκής συνεργασίας στην επιβολή του νόμου, δηλαδή μεταξύ των, των ε, μέτρων κατά της εγκληματικότητα. Αυτό προκαλεί μια σχετική ένταση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το παραβλέψουμε. Uh, Εδώ φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα το ζήτημα αυτό, η μέρημνα αυτή. Είναι λοιπόν ε, αναπόφευκτο να λάβουμε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτήν την ένταση που επικρατεί και να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία. Το δεύτερο σημείο τώρα είναι ότι ο τομέας αυτός ε, εξελίσσεται διαρκώς και με γοργούς ρυθμούς. Κανείς πριν από 20 χρόνια δεν θα μπορούσε να μαντέψει ότι σήμερα θα φτάναμε σε αυτό το σημείο ως προς την επικοινωνία, τη μεταφορά δεδομένων και ούτω καθεξής. Ε, Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαι πλήρως πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικαιροποιήσει την προηγούμενη νομοθεσία της. Για προφανείς λόγους πρέπει να είναι ε, να λάβει υπόψη και να καλύψει τις σημερινές ανάγκες. Και αυτό ίσως να κάνει κάποιους να αισθάνονται άβολα, αλλά το θέμα αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον αναγκαστικά ίσως να πρέπει να το ξαναδούμε θα επανέρχεται διαρκώς και νομίζω ότι θα καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβαλλόμενη, διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τον τρόπο που θα προστατεύονται και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν η συζήτηση αυτή ε, είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και πλούσια. Ελπίζω να τη βρίσκουν ε, το ίδιο χρήσιμη και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων όπως και το Ευρωκοινοβούλιο και θα ενώσω τη φωνή μου με αυτούς που λένε ότι σε, στην πράξη είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ διεθνούς χαρακτήρα και εθνικού χαρακτήρα δεδομένων. Οι δέσμοι μέτρων, όπως προτείνεται, το πακέτο αυτών των προτάσεων, ε, σαφώς χρήζουν τροποποιήσεων και προσαρμογών, ώστε να λάβουμε υπόψη τα δύο άκρα της, ε, της έντασης που έχει δημιουργηθεί, αλλά Σίγουρα πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία ψηφιακή αγορά που όλοι επιδιώκουμε και θα είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό για την μελλοντική ανάπτυξη των ε, οικονομιών μας. Ευχαριστώ. Και με τη σειρά τώρα δίνω το λόγο στην Ταϊάννα Αλόνσο Μπλάς τα θέματα διαφάνειας, εμπιστοσύνης και επαγγελματικών ε, υπευθύνων. Ευχαριστώ πολύ και μετά από τις παρεμβάσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων, ιδίως μετά από σεφή η Άννα εδώ στα αριστερά, νομίζω ότι το σύστημά μα ε, προσφέρει ψηλότερη προστασία από την προτινόμενη οδηγία και μήπω είναι καλύτερα να παραμείνουμε σε αυτό. Είναι ένα θέμα αλλά έθεσε κάποια ζητήματα και ο κύριος Άλβαρο για την ακρίβεια των ε, δεδομένων και θέλω να απαντήσω σε αυτό. Είναι θεμελιώδους σημασία σε αυτό. Είναι ένα από τα λίγα ζητήματα όπου οι υπεύθυνοι της προστασίας δεδομένων αλλά και οι υπεύθυνοι υποβουλής του νόμου συμφωνούν. Είναι ζωτική σημασία να είναι ε, ακριβή τα δεδομένα. Να μην ε, συλληφθεί, για παράδειγμα, λάθο άνθρωπο βάσει λανθασμένων πληροφοριών. Βεβαίω, αυτό είναι κυρία σημασία. Όταν βεβαίω κανεί εργάζεται, σε διεθνέ πλαίσιο, είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Οι πληροφορίε προέρχονται από διαφορετικέ πηγέ, όπω τι δικαστικέ αρχέ διαφορετικών χωρών. Αυτό που σε κάθε περίπτωση έχουμε προβλέψει και λειτουργεί αποτελεσματικά είναι ένα σύστημα όπου οι πληροφορίε ε, συγκρίνονται μεταξύ των υπευθύνων για τη διαχείριση τη κάθε υπόθεση και μόλι προκύψουν διαφορέ μεταξύ των πληροφοριών από διαφορετικέ πηγέ, τότε τι αντιπαραβάλλουμε για να γίνει επαλήθευση. Έπειτα υπάρχει ένα αρχείο μεταφορά των δεδομένων, οπότε ο καθένα που έχει αποστείλει μια πληροφορία ε, γνωρίζει τι συνέβη και σε ποιον κατέληξε η πληροφορία. Αυτό λοιπόν με το τεχνικό μα σύστημα είναι πολύ απλό να γίνει, γιατί καταγράφουμε ακριβώ και την πηγή και τον παραλήπτη τη πληροφορία. Είναι εξαιρετική σημασία στο στοιχείο αυτό. Ω προ τα σχόλια τη κυρία Σίπελ. Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω και να επιρώσω τα όσα είπατε, διότι η εμπιστοσύνη είναι καθοριστική σημασία. Βεβαίω για τον κύριο Τζαστ αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι εθνικέ αρχέ μα εμπιστεύονται. Ότι συνειδητοποιούν ότι το σύστημα προστασία δεδομένων που διαθέτουμε είναι επαρκέ. Εδώ ε, εξαρτώμαστε ε, από τις εθνικού ανακριτέ, του εθνικού αρμοδίου που φέρνουν σε εμά τι υποθέσει. Από αυτό εξαρτάται η λειτουργία μας. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήταν πολύ σημαντικό να ισχύσει κάτι ανάλογο και σε εθνικό επίπεδο. Δείτε, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, έχει πολύ διαφορετικές υποδιαγραφές για τις ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες που ασχολούνται με την ε, επιβολή του νόμου από ό,τι ισχύει σε εθνικό. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε, διότι το νομικό μας σύστημα δεν θα μας το επέτρεπε. Αυτά μπορούν να γίνουν απλά μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό ισχύει και για το τι προκύπτει από τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα σε τρίτες χώρες εάν δεν υπάρχουν ανάλογες συμφωνίες, αν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις. Για την ώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα στι περισσότερε υποθέσει. Υπάρχουν κάποιε φορέ διμερεί συμφωνίε με ασάφειε, αλλά πολλέ φορέ τα πράγματα αυτά ε, γίνεται να επιληθούν. Είναι ε, μια πολύ καλή ε, ευκαιρία να τα δούμε τα πράγματα από μια ευρύτερη σκοπιά. Σα ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκρέβερ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγιναν πολλές ε, εύστοχες παρατηρήσεις και απευθύνθηκαν κάποιες ερωτήσεις και σε εμάς. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω κάποιες σύντομες απαντήσεις. Όταν μιλάμε για την πρόσβαση των δικτικών αρχών σε δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, αλλά από ιδιωτικές πηγές, και βεβαίως βλέποντας τα πράγματα από τη σκοπιά της Europol, ε, να σας πω ποιο σύστημα έχουμε εμείς στη Europol. Η Europol δεν έχει τη δυνατότητα απευθείας να απευθυνθεί σε ιδιωτικέ εταιρείε και να του ζητήσει δεδομένα. Έχουμε όμως ένα σύστημα με εχέγγυα για την προστασία των δεδομένων και εφόσον τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη τρομοκρατία, τότε μπορεί να μα να παρασχεθούν από τι εθνικέ αστυνομικέ αρχέ, οι οποίε αποκτούν τα δεδομένα αυτά βάσει των εθνικών διαδικασιών που προβλέπει το δίκαιο τη χώρα του δηλαδή. Αυτά θα επηρεαστούν φυσικά και από την οδηγία που συζητούμε εφόσον εγκριθεί. Αναφέρατε και τη διαφάνεια. Η διαφάνεια ε, για τη Europol και την υπηρεσία μας είναι Κάτι το σημαντικό προφανώς, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθεία στην υπηρεσία μας, όχι μόνο για να επιθούν ε, ε, δεδομένα και την πρόσβαση σε αυτά, αλλά και για πληροφορίες ανάλογα με τα έγγραφα που εμείς δημοσιοποιούμε. Από την πλευρά λοιπόν της λογοδοσίας και επειδή είμαστε υπηρεσία επιβολής του νόμου, ε, πρέπει να λογοδοτούμε και για το αστυνομικό έργο που διεξάγουμε. Επίσης, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό για την ε, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνη ε, με του Ευρωπαίου πολίτε και προς τι ε, αρχέ επιβολή του νόμου. Ειδικά για την Europol όμως. Εάν τα κράτη-μέλη, οι εθνικέ αστυνομικέ αρχές δεν εμπιστεύονται την Europol ότι έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί τα δεδομένα ως ένα κομβικό σημείο διαχείρισης των δεδομένων αυτών. Και ότι συμμορφωνόμαστε με τους αυστηρότατους κανόνες προστασίας δεδομένων, τότε θα σταματήσουν οι ροές πληροφοριών προς εμάς. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι εγγύησεις και εφόσον οι διαδικασίες δεν είναι νόμιμες, δεν θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε τελικά ε, ως αρχή. Εκεί λοιπόν έρχονται και συναντώνται τα συμφέροντα και οι ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, ε, οι ανάγκες συλλογής των δεδομένων και βεβαίως όλα αυτά να ε, τα επεξεργαζόμαστε με βάση τους ισχύοντες κανόνες. Χρειάζονται ακριβή και υψηλή ποιότητα δεδομένα στι βάσει δεδομένων μα. Αυτό χρειάζονται οι διοικητικέ αρχέ. Και από αυτή τη σκοπιά, οι κανόνε για την προστασία των δεδομένων, τη Europol, και αν δείτε τι λεπτομέρειε των κανόνων ακριβώ, ε, έχουμε πλήρη ε, καταγραφή των δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την ε, συλλογή και την τήρηση ανάλογων αρχείων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη δική μου πλευρά ένα μόνο σχόλιο, διότι εκπροσωπώ το επιχειρησιακό σκέλος της Europol να επικεντρωθώ στις πρακτικές διαστάσεις της επιβολής του νόμου και τα όσα συζητήθηκαν. Από αυτό που ανέφερε και η Ζήπελ, για τους διαφορετικούς τρόπους επεξεργασία ή αποστολή πληροφοριών μεταξύ των κρατών Αυτή την πρόκληση την έχει αντιμετωπίσει η Europol, ιδίω στην αρχή της λειτουργία της. Υπάρχει νομοθετική πράξη που επιτρέπει την ε, ε, παραλαβή και αποστολή πληροφοριών. Χρειάστηκε βέβαια να ευαισθητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη, να τα ενημερώσουμε και να του εξηγήσουμε ποια είναι τα κριτήρια που ισχύουν για μα. Πώ ε, πρέπει να είναι τα δεδομένα για να τα αποδεχτούμε στην Europol. Και οι πληροφορίε που αποστέλνουμε εμεί στην Europol. Εδώ θα έρθω και στα σχόλια που έκανε ο η κυρία Μπούσερ, για την ε, επεξεργασία των δεδομένων. Η προπόθεση αυτή είναι απαραίτητη ε, και πρέπει να αποδεικνύεται η, χρησιμο... η αναγκαιότητα του σκοπού προκειμένου να αποδεχτούμε εμείς μια πληροφορία. Δηλαδή εμείς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μας για την καταπολέμηση του δεδομένου εγκλήματος. Και μπορεί ανα πάσα στιγμή ο καθένα να μα ε, ρωτήσει γιατί τα δεδομένα αυτού του ατόμου τα έχετε στο σύστημά σα, γιατί τα επεξεργαστήκατε, γιατί τα διατηρήσατε για τόση χρονική διάρκεια. Ποιο σκοπό εξυπηρετούσε η τήρηση των ε, δεδομένων αυτών στο σύστημά σα. Έτσι λοιπόν Έχουμε προσπαθήσει σκληρά για να είναι σκόπιμε πληροφορίε που συγκεντρώνουμε και το αποδέχονται όλε οι αστυνομικέ αρχέ με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Και στα κάτι μέλη ιδιοκτικέ αρχέ κατανοούν ότι υπάρχει ανάγκη εναρμόνιση. Θα διευκολυνθεί το έργο τη αστυνομία εάν ο αστυνομικό ξέρει ποιοι είναι οι κανόνε του παιχνιδιού όταν αποστέλει πληροφορίε σε μια άλλη χώρα. Και πώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίε αυτέ. Διότι τελικά η επεξεργασία των ε, δεδομένων δεν γίνονται για τη χαρά τη επεξεργασία. Πρέπει να τα αποστείλουμε ξανά στα κρατημέλη και τέλο πάντων ο απότερο σκοπό είναι να υπάρχει πρόσβαση με... Ε, και δυνατότητα επιβολή ποινών. Καταδίκη. Ε, αυτό είναι ο στόχο του νόμου. Ευχαριστούμε. Και δίνω το λόγο στην κυρία Έλση Um, one... Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω να κάνω ως προς τις παρατηρήσεις του κυρίου Άλβαρο. Συμφωνώ για το περιορισμό του σκοπού και για τα άλλα πρότυπα της προστασίας δεδομένων. Ήταν ήδη προβληματικά όλα αυτά στη Συμφωνία Πλαίσιο. Περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί και εκείνοι αναθεωρούν τα δικά τους κείμενα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν ιδιαίτερω τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων. σω κάποιε λεπτομερίες αλλάξουν και αυτό κάνουμε και εμεί άλλωστε σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το τοπίο του επόμενου μήνε. Τώρα, ω προ την πρόσβαση των αρχών επιβολή του νόμου στι πληροφορίε και στα προσωπικά δεδομένα από ιδιωτικέ επιχειρήσει, και εδώ θέλω να τονίσω το προαπαιτούμενο της αναγκαιότητας που ε, ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής. Εάν πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει ένα τόσο μη συμβατό ε, σκοπό, τότε η αρχή της αναγκαιότητας είναι η μόνη λύση, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη η συζήτηση αυτή. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν θέλουμε να ξαναγίνει συζήτηση που είχαμε με τη συμφωνία SWIFT, με το πρόγραμμα ε, ανείχνευσης και ειχνηλασιμότητας για ε, θέματα τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε ε, τη συζήτηση που έγινε για τις υπηρεσίες και επιχειρήσεις ψαρέματος. Πράγματα δηλαδή που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ιάννα. Θέλω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσαν οι συμμετέχοντες. Πρώτον, το θέμα της διαφάνειας. Πολύ σημαντικό. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω τη διαφορά μεταξύ του κανονισμού και της οδηγίας. Ο κανονισμός στο άρθρο 5α, θεμελιώδεις αρχές, δίκαιη επεξεργασία, απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων με διαφανή τρόπο. Η οδηγία δεν το, δεν το κάνει αυτό. Στο άρθρο 4α αναφέρεται η δίκαιη επεξεργασία και δεν γίνεται καμία μνήμα στην διαφάνεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι Πράγματι, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένε περιπτώσει στι αρχέ επιβολή του νόμου όταν αυτέ δραστηριοποιούνται. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε μια παρέκκληση του στυλ όπου δει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπάρχει διαφάνεια σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό υποθέσεων με τις οποίες ασχολούνται οι αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό καταρχάς για το θέμα της διαφάνειας. Από εκεί και πέρα, αναφερθήκατε στην εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι και ο λόγος άλλωστε που όταν πήρα το λόγο προηγουμένως είπα ότι είναι πολύ σημαντικό εάν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δουλεύουν πάνω σε έναν κοινό οδικό χάρτη για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων, εκεί θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα πάντα, από τη μετάφραση προς την, μέχρι και την πρόσβαση. Να μην είναι αποκλεισμένα τα δεδομένα και η προστασία Του Είναι γελίο αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει στον οδικό χάρτη αναφορά στην προστασία των δεδομένων. Είδα αλλιώ θα καταλήξουμε να έχουμε ισχυρότερες διατάξεις στο χ κράτος μέλος και πιο δύναμε διατάξεις στο ψ κράτος μέλος. Πώς θα πετύχουμε την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων. Και αυτό με φέρνει πάλι σε αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή ο κατακαιρματισμός. Η κυρία Ρέντιν ανέφερε ότι σκοπός του πακέτου αυτού είναι η απλούστευση και η έλλειψη κατακαιρματισμού. Δεν πρόκειται όμως τελικά να διαπιστώσουμε έλλειψη κατακαιρματισμού πέρα από τα 27 διαφορετικά καθεστώτα, κανόνες για τις αρχές επιβολής του νόμου, έχουμε την οδηγία για την ιδιωτικότητα, για την διακράτηση των δεδομένων, επίσης την οδηγία. Όλα αυτά αναφέρονται στην προστασία των δεδομένων. Πώς γίνεται να έχουμε απλούστευση όταν έχουμε τρεις διαφορετικές οδηγίες κτλ. Ε, θα πρέπει να τα δουλέψουμε όλα αυτά κάπως περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι κλείσαμε την τρίτη συνεδρία και σας ευχαριστώ όλους εσάς ε, που ήσασταν κοντά μου εδώ στο πάνελ. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις σας. μπορούμε με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το προς τα που θα κινηθούμε στο μέλλον. Πήγαμε, πήραμε και πρακτικά στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ όλους και για την προσοχή σας και τηρήσαμε και το χρόνο που μας είχε δοθεί. Και τώρα θα ζητήσω από τους συναδέλφους Νάντια Χίρς και Σον Κέλλη να έρθουν να αναλάβουν το συντονισμό της τέταρτης συνεδρίας. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η τέταρτη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.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 Members, uh, national parliamentarians, ladies and gentlemen. Ε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, αγαπητοί φίλοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φτάνουμε στην τελευταία συνεδρία ε, της σημερινής μας ημέρας και ίσως και την πιο σημαντική. Πριν, είναι η δεύτερη φορά που μου δίνουν τέτοιο σφυράκι σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και θα το χρησιμοποιήσω όσο και όπως μπορώ. Σας ενημερώνω. Χαίρομαι διότι είμαι συγητής της Επιτροπής Ήτρε για αυτή την πολύ σημαντική πρόταση. Τους τελευταίους μήνες έχω συναντηθεί με πάνω από 120 ομάδες άσκησης, πίεσης και συμφερόντων με διάφορα λόμπι που μου έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τις προτάσεις. Γενικότερα ε, υπάρχει θερμή υποδοχή και ελπίζουμε όλοι ότι θα καταλήξουμε σε έναν καλό κανονισμό. Θα μιλήσουμε για τη συγκατάθεση, για τη ρητή συγκατάθεση, για την ε, λανθάνουσα συγκατάθεση, για το δικαίωμα στη ψηφιακή λύθη, για το online, το offline, το PPO για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων και για τις γνωστοποιήσεις και το καθεξής. Θα συζητήσουμε λοιπόν κάτι το πολλά και σημαντικά πράγματα. Εκτελούνται στην επεξεργασία δεδομένων και υπεύθυνοι τη επεξεργασία δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα και στον τομέα τη απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό να τα πάμε καλά σε αυτό το επίπεδο, να, γράψουμε τα σωστά πράγματα στα νομοθετήματα τελικά. Να υπάρχει λογοδοσία κατά κύριο λόγο του ελεκτή, εάν αγοράσει κανείς ένα αυτοκίνητο και χαλάσουν τα φρένα, δεν ε, ζητάει τα αρέστα από το εργοστάσιο που κατασκεύασε τα, φρένα, πηγαίνει κατευθείαν στην αντιπροσωπεία από όπου αγόρασε το αυτοκίνητο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει λογοδοσία γενικότερα. Και για να χρησιμοποιήσουμε πάλι αυτή τη μεταφορά των αυτοκινήτων, το, θα έλεγα ότι πράγματι ε, ε, εδώ έχουμε την εποχή της ψηφιακής αυτοκίνησης. Δηλαδή τώρα θεσπίζουμε και φτιάχνουμε ένα κώδικα όχι οδικής κυκλοφορίας αλλά ψηφιακής κυκλοφορίας. Τους κανόνες με τους οποίους όλοι ε, θα οδηγούμε και θα πλοηγούμαστε σε αυτό το ψηφιακό κόσμο. Και νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε σωστή δουλειά και ότι ο κανονισμός στον οποίο θα καταλήξουμε το 2013-2014 θα αντέξει στο χρόνο ε, στρέφομαι στην ε, εξαίρετη συνάδελφο που κάθεται εξ αριστερών μου, την ε, κυρία Νάντια Χίρς και της δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ως συντονίστρια εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης, γιατί εγώ ανέλαβα τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, και ασχολήθηκα με το θέμα της προστασίας δεδομένων είναι θέματα τα οποία αναγράφονται στο άρθρο 82 όσον αφορά την, τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων στις επιχειρήσεις. Υπάρχει εκπροσώπηση εργαζομένων και συνδικάτων και στην αρχή δεν ε, το είχαμε σκεφτεί ότι η προστασία δεδομένων αφορούν ε, τους εργαζομένους, όμως σιγά σιγά ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους και τα συνδικάτα και έχουν προκύψει και διάφορα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο προέκυψε είναι ότι ε, στα, κράτη, στα διάφορα κράτη-μέλη ακολουθούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι γίνεται με τα δεδομένα. Και πριν από 10 χρόνια είχε γίνει μια αρχική προσπάθεια της Επιτροπής να βρεθεί μια κοινή γραμμή, αλλά απέτυχε, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο τομέας. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία των ε, εργαζομένων και τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες ε, σε αυτόν τον ε, τομέα υπάρχουν καταχρήσεις των δεδομένων των εργαζομένων έχουν τύχει περιστατικά όπου κατεγράφησαν και με οπτικοακουστικά μέσα ε, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Έχει συζητηθεί λοιπόν πάρα πολύ το θέμα. Το άρθρο 82 είναι το βασικό άρθρο που ενδιαφέρει την Επιτροπή Απασχόλησης και τους εργαζομένους γενικότερα και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια θέματα που προχωρούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή ότι θέλουμε να υπάρχει ε, δυνατότητα για τα κράτη-μέλη ε, να εφαρμόζουν την εθνική τους πολιτική, αλλά να υπάρχουν και κάποια ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να αποδέχονται όλα τα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη, ένα σημείο που λέει ότι οι εργαζόμενοι ε, έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται από τον εργοδότη για το ποια δεδομένα έχουν αποθηκευθεί, ποια προσωπικά τους δεδομένα ε, τηρούνται και θα πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ε, πόσα δεδομένα δίδονται στις, τηλε... εταιρείε τηλεπικοινωνιών, ε, πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των ε, ηλεκ... μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία της περιαγωγής, κατά πόσο λαμβάνονται, κατά πόσο καταγράφονται και διατηρούνται όπως επίσης το δικαίωμα στο να μην γίνεται βιντεοσκόπηση χωρίς την αδειά τους. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι σημαντικό το να ξέρουμε αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μέσα στην επιχείρηση και πότε γίνεται αυτό και μία από τις βασικότερες απαιτήσεις ε, είναι νομίζω το θέμα της έλλειψης ισορροπίας ε, μεταξύ ε, εργοδοτών και εργαζομένων, διότι είναι διαφορετικό το επίπεδο εξουσίας που υπάρχει και πολύ συχνά το έχουμε συζητήσει με εκπροσώπους των εργαζομένων ότι πολλές φορές προσφέρονται στους εργαζομένους κάποιες πρόσθετες παροχές όπως ασφαλιστικές παροχές παραδείγματος χάρη σε αντάλλαγμα με την παροχή κάποιων δεδομένων και πρέπει να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι, εφαρμόζονται οι αρχές του να είναι επωφελές αυτό για τους εργαζομένους. Χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και που συμμετέχω και στο Προεδρείο Συντονίστρια και θα έλεγα να ξεκινήσουμε κατευθείαν ε, με τον συνάδελφο εξ αριστερών, τον συνάδελφο από την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Στέφαν Μάγερ. Καλώς ήρθατε και σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να συζητήσουμε αυτό το δύσκολο θέμα και πολύ φιλόδοξο θέμα για την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ένα κεντρικό σημείο των προσπαθειών της Επιτροπής που έχει συζητηθεί και στο παρελθόν. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται δημοσίως ε, ε, και στην κοινή γνώμη αλλά και στο, στη Γερμανική Βουλή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη Γερμανία. Η οικονομία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ως ε, νόμισμα. Δεν είναι το κράτος που τα χρησιμοποιεί, αλλά η οικονομία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια κατευθυντήρια γραμμή που να σταθμίζει και τα συμφέροντα των εργαζομένων και τα συμφέροντα αυτών που χρησιμοποιούν τα δεδομένα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν είναι μεμονωμένο. Υπάρχουν και τα άρθρα 15 και 16 που επίσης ε, είναι άρθρα της, ε, του Χάρτη Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πολλές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων εξετάζονται από την πλευρά των ε, καταναλωτών. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν διατάξεις ε, για ε, την ιδιωτικότητα βάσει σχεδιασμού και την ιδιωτικότητα βάση ρυθμίσεων που βρίσκονται εξ αρχής μέσα στο σύστημα και αυτά είναι αυτά τα οποία λαμβάνονται υπόψη, αυτά τα οποία κατασκευάζονται στο, στις υπηρεσίες διαδικτύου. Ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τη γραφειοκρατία και να μειώσει και το κόστος για τις επιχειρήσεις νομίζω ότι δεν επιτυγχάνεται με αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν υποχρεώσεις παροχής δεδομένων το άρθρο 14 και 15 και το άρθρο 32 ε, ε, περιλαμβάνουν πολλές απαιτήσει δεδομένων και δεν είναι σαφές ποια υποχρέωση παροχής δεδομένων ε, έχουν οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν θέματα στα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση παροχής πληροφοριών και θα μπορούσα να το διευκρινίσω αυτό. οι πληροφορίες που υπάρχουν σε επιχειρηματικές κάρτες θα μπορούσαν να αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από τις ε, επιχειρήσεις και πολλές από τις νέες απαιτήσει είναι απαιτήσει οι οποίες μεταφέρονται στις ε, επιχειρήσεις. Από αυτό θα πλήττονται ε, ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις που θα πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό περιθώριο 24 ωρών να μπορούν να δώσουν διευκρινήσεις για οποιασδήποτε πληροφορίες λυθούν σχετικά με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει ένα όριο ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει το όριο των 250 εργαζομένων για να μπορεί να υπάρχει αντίστοιχη προστασία δεδομένων. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση των υπηρεσιών προστασίας δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Υπάρχει η νέα αρχή της μονοαπευθυντικής ε, θηρίδας. Ακόμη και αν ισχύσει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο η έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερε ρυθμίσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ και πολλά χρόνια στην Γερμανία υπάρχουν πολλοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων σχετικά με τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και νομίζω ότι και εδώ έχει πολλά ακόμη να κάνει η οδηγία ή ο κανονισμό για να καλύπτει τα θέματα των δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις. Ε, υπάρχουν συμφωνίες μέσα στις επιχειρήσεις σχετικά και με τα δικαιώματα των εργαζομένων και η διαδικασία της υποβολής δεδομένων και η διαδικασία της συλλογής δεδομένων είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο άρθρο 6, 1, β και γ σχετικά με την παροχή δεδομένων στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υποχρέωσης. στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασία στη Γερμανία υπάρχουν αντίστοιχε ρυθμίσει για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, στο άρθρο 7, παράγραφος 4, υπάρχει το θέμα της συγκατάθεσης ε, σε ε, σχέση και με το άρθρο 34 και αναφέρεται ότι όταν είναι εξαρτημένη η σχέση εργασία με τον υπεύθυνο προστασία δεδομένων μέσα σε μια επιχείρηση όταν μιλάμε για εργαζομένου, υπάρχει, ε, ακυρώνεται αυτή η ε, εξαίρεση της συγκατάθεσης. Όταν προσφέρονται επιπλέον ασφαλιστικές προσφορές από τον ε, εργοδότη προς τους εργαζομένους και πάλι υπάρχουν θέματα προσωπικών δεδομένων τα οποία ε, δίδονται στην επιχείρηση στο πλαίσιο των ε, ασφαλιστικών υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν και θα πρέπει και αυτά, να, αυτά τα στοιχεία να υπόκειται στην προστασία των δεδομένων. Όσον αφορά τις πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση, θα ήθελα επίσης ε, να πω δύο λόγια. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα σημεία, πάνω από 50 σημεία που υπάρχουν ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση και υπερβαίνουν αυτά τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 290 της συνθήκης σχετικά με τις δυνατότητες της Επιτροπής ε, να θεσπίζει πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Το σχέδιο κανονισμού δεν προβλέπει μόνο συγκεκριμένα σημεία, αλλά ε, προβλέπει και τη δυνατότητα της Επιτροπής ε, να παρεκκλίνει από αυτές τις διατάξεις. Θα έχει λοιπόν η Επιτροπή τη δυνατότητα να θεσπίζει μόνη της κάποια σημεία τα οποία θα έπρεπε να θεσπίζονται από τον κανονισμό. Ο αριθμός των πράξεων κατεξουσιοδότηση κατά τη γνώμη μου πρέπει να μειωθεί κατά πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία κατά τους προσεχείς μήνες και εβδομάδες να καλύψουμε αυτά τα θέματα και να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωσή τους. Θα πρέπει να προβλέπετε συνεκτικότητα στον κανονισμό και για λόγους κράτους δικαίου. οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα πρέπει να συνεχίζουν να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες παράλληλα με την προστασία δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι η διαδικασία που προβλέπεται ε, για τις Εθνικές Αρχές Δεδομένων ε, δεν ε, συμβαδίζουν με το άρθρο 20 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την αρχή της, για τις δημοκρατικές αρχές. Στις συζητήσεις στη Γερμανία εξετάζουμε τα θέματα της πρακτικής εφαρμογής των ε, διατάξεων αυτών και η συζήτηση θα συνεχιστεί. Συζητείται και το θέμα ε, των αγωγών από συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, από σωματεία ή και η άσκηση συλλογικής ε, αγωγής. και για πολλούς ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνέπειες από τον ε, κανονισμό αυτό. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ένα νομοθετικό κείμενο που δεν έχει πρακτικές επιπτώσεις στις ζωές των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ, Στίβεν, και σε ευχαριστούμε διότι δεν ξεπέρασες το χρόνο σου. Παρόλο που ε, με αυτό το ρυθμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να σε ακολουθήσουν οι διερμηνείς. Και θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον διερμηνέα που σε διερμήνευε από τα γερμανικά προς τα αγγλικά γιατί πράγματι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια. Προχωρούμε τώρα στην κυρία Έρικα Μαν, μια πολύ ισχυρή κυρία, γενική διευθύντρια του Facebook και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Μαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για, την, ε, για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και για το ότι μας καλέσατε εμάς στο Facebook να συμμετάσχουμε στις συζητήσεις σας. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις πριν αναφερθώ στο ερωτηματολόγιο σας. Η αναθεώρηση της οδηγίας και του κανονισμού πράγματι μπορεί να διευκολύνει την καινοτομία και συνάμα να προσφέρει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο του διαδικτύου. Το Facebook πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε και κανονισμό για την ιδιωτικότητα και ανθίζουσα ε, διαδικτυακή σφαίρα. η διαφάνεια, ο έλεγχος, η λογοδεσία αντιστοιχούν στα μέτρα που υπάρχουν ε, στον κανονισμό για την ιδιωτικότητα και για την, των δεδομένων. Τώρα, η μείωση του ρυθμιστικού και διοικητικού άγχους για τους controllers, για τους ε, εκτελούντες στην επεξεργασία ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή για κάθε επιχείρηση που απασχολεί άνω των 250 εργαζομένων θέλει να υπάρχει θέση ατόμου που διαχειρίζεται αυτό το θέμα. Και σε κάθε περίπτωση το διοικητικό άχθος και το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλο. Όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις. Το Facebook καταλαβαίνει τις δυσκολίες της Κομισιόν, ε, του Κοινοβουλίου πόσο δύσκολο είναι να βρούμε ένα σημείο ισορροπία μεταξύ της ε, τη της ανάκαψης και της ύπαρξης ε, εγγυήσεων για τα προσωπικά δεδομένα. Είμαστε σε ένα πρωταρχικό ε, στάδιο της ανάπτυξης του διαδικτύου. Νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε φτάσει στο τέλος, όμως όχι, είμαστε στην αρχή ως προς το διαδίκτυο. Επιχειρήσεις, οι ιδέες εξελίσσονται, αλλάζουν και θα πρέπει η νομοθεσία να μην ε, αποτελεί ένα περαιτέρω επιπρόσθετο βάρος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, είτε τις μικρομεσαίες είτε τις μεγαλύτερες. Το 2010 η Κομισιόν αναγνώρισε τη σημασία του ψηφιακού τομέα, του διαδικτυακού τομέα στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη έχουν συχνά εκφράσει την πίστη τους στην ψηφιακή οικονομία, η οποία θα μπορέσει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δραστηριοποιούνται δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία και οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις παγκοσμίω είναι ευρωπαϊκές. Η Skype από το ε, Λουξεμβούργο, Visa Γαλλία, ε, Book από τη Γερμανία. Πάρα πολλές επιχειρήσεις που ανθούν στο ψηφιακό κόσμο είναι ευρωπαϊκές. Στα επόμενα χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία θα είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το Facebook έχει τύχει να συνεργάζεται με αυτές τις startup, με αυτές τις ψηφιακές εταιρείες. Έχουμε μεγάλη αισιοδοξία για την ποιότητα και τη δημιουργικότητα όλων αυτών των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά μόνο, ε, τις startup και πιστεύουμε ότι θα προσεγγίσουν πάρα πολλούς χρήστες και καταναλωτές παντού. Η Deloitte ε, στη μελέτη της δείχνει ότι από τις δραστηριότητες του Facebook στην Ευρώπη ε, η αξία αυτή μεταφράζεται σε 32 δις. Και νομίζουμε ότι έτσι, βάσει της έρευνας της Deloitte, ε, ενισχύθηκε η δημιουργία άνω των 230.000 θέσεων απασχόλησης. Τώρα, ω ως, ως προς το ε, πώς η μονοαπευθυντική θηρίδα του One Stop Shop θα επηρεάσει την εθνική νομοθεσία, πώς θα ε, είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο ε, θα ε, είναι ομοιόμορφες και δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού του μηχανισμού. Θα υπάρξει περισσότερη εναρμόνιση στην νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και θα υπάρξει μεγαλύτερη νομική ε, εναρμόνιση ως προς τη δικαιοδοσία για την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων και έτσι θα μειωθεί και το κόστος που προκύπτει από, τις, από τα διαφορετικά καθεστώτα ανά την Ευρώπη. Θα διευκολύνουμε έτσι την προστασία και την ροή των δεδομένων μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Να επανέλθουν συντομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο ψηφιακό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα είναι κλειδί για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αρχή της μοναπευθυντικής θηρίδας θα ενισχύσει την τάση αυτή. Τα στοιχεία της Deloitte είναι πολύ εύγλωτα. Θα σας μιλήσω για έναν άλλο αριθμό από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής, το οποίο έχει βρει ότι, για παράδειγμα, Μία ολοκληρωμένη ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά θα είχε αύξηση ΑΕΠ κατά 4%, δηλαδή 500 δις ευρώ σε μία περίοδο 10 ετών. Αυτή είναι η εκτίμηση. Πρέπει κανείς βέβαια να είναι προσεκτικός με αυτούς τους αριθμούς γιατί οι αριθμοί εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί τελικά η ευρωπαϊκή οικονομία και πώς θα εξελιχθούν και θα λειτουργήσουν τελικά οι αγορές παγκοσμίως. Αλλά εν πάση είναι ενδιαφέροντα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Ο μηχανισμός το One Stop Shop της μονοαπευθυντικής θηρίδας είναι ένας μηχανισμός που θα πρέπει να αφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις καινοτόμε επιχειρήσεις για να ανθίσουν, να μην έχουμε κατακαιρματισμό, να μην έχουμε επιπρόσθετο διοικητικό βάρος. Άλλωστε η Κομισιόν έχει αξιολογήσει ότι 2,2 ευρώ, έχει εκτιμήσει ότι 2,2 ευρώ είναι το λογαριασμός για το διοικητικό βάρος ανά έτος. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες για επενδύσεις στην Ευρώπη και αυτός ο μηχανισμός θα λειτουργήσει μόνο εάν η σχέση μεταξύ εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και ε, της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία έχει σχέση με το που εδρεύει η επιχείρηση, ε, καθορίζεται πλήρως η σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Στο σχέδιο κανονισμού έχουμε μια σειρά άρθρων που μπορούν να υπονομεύσουν την ε, εξουσία του DPA μπορεί τελικά να ε, ε, επιδεχθεί διαφόρων ερμηδινιών το προβλεπόμενο και η διατύπωση εκεί αναϋπόθεση, αναπερίπτωση. Και είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να το εξετάσει αυτό εκ του να υπάρχει συνοχή δηλαδή μεταξύ όλων αυτών των διατάξεων ε, συνοχή μεταξύ των ορισμών και ενδεχομένω θα μπορούσαν να υπάρξουν και συστάσεις Τώρα, ως προς το Facebook, εμείς έχουμε την έδρα μας στην Ιρλανδία από το 2010, άρα υποκείμεθα στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας, τον DPC δηλαδή, εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, συμμορφωνόμαστε και τις στηρούμε ως προς την ιδιωτικότητα. Έχουμε στενή συνεργασία όπου δει και όπου μπορούμε με την αρχή, την Ιρλανδική για την προστασία των δεδομένων. Το Facebook πρόσφατα υπέστη ενδελεχή έλεγχο από την αρμόδια Ατλαντική Αρχή για την ιδιωτική σφαίρα, για την ιδιωτικότητα και να σας πω ότι για τρεις μήνες μας εξέτασαν ενδελεχώς και συνέταξαν την τελική τους έκθεση στην οποία αναφέρουν ότι όχι μόνο συμμορφωνόμαστε πλήρως με την Ιρλανδική νομοθεσία αλλά έχουμε υιοθετήσει και τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την προστασία των δεδομένων. Μετά από τρεις μήνες ερευνών η έκθεση ήταν ξεκάθαρη υπερημών και μετά είχαμε έξι μήνες κοινή εφαρμογής. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο, η Ιρλανδική αρχή ε, στην έκθεσή της επανέλαβε ότι το Facebook έχει ε, ε, εκφράσει πάγια δέσμευση να συμμορφωθεί με τα ε, επιβαλόμενα. Μας μένουν λίγες εβδομάδες για να κάνουμε κάποιες αλλαγές, δεν έχει λήξει ακόμα αυτή η προθεσμία και ε, βεβαίως θα τηρήσουμε τις ε, δεσμεύσεις μας εντός ε, της οριστής σας προθεσμίας. Και τέλος, θέλω να αναφερθώ στο εξή ερώτημα. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι αυτό το σχέδιο κανονισμού και σχέδιο ε, οδηγίας θα ε, ε, είναι στο ύψος των τεχνολογικών εξελίξεων, δηλαδή θα ακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η τεχνολογία. Εμείς είμαστε υπέρ της αρχής by design, από σχεδιασμό και όχι της αρχής by default, εξορισμού. Ενδεχομένως το εξορισμού δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση των δικτύων ε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλοι θέλουν να μοιράζονται και να συνδέονται με τους άλλους. Το μοιράζομαι και το συνδέομαι είναι και ο πυρήνας αυτού του ψηφιακού προϊόντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποκτά κανείς λογαριασμό στο Facebook, γιατί θέλει να μοιράζεται και να συνδέεται. Ε, γι' αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει το site μας έτσι ώστε να ελέγχουν οι καταναλωτές, οι χρήστες μάλλον, με, το, ποιους θα μοιράζονται το περιεχόμενο που θέλουν να μοιράζονται. Ε, και τον έλεγχο αυτό τον υποστηρίζουμε με πολύ απλά εργαλεία στα οποία δίνουμε, για τα οποία δίνουμε πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Μπορούν να κατεβάσουν τα δεδομένα και να ελέγξουν τι δεδομένα ήδη έχουν ε, βάλει στο Facebook. Μπορούν εύκολα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις για την ιδιωτικότητα και το Facebook επίσης πιστεύει ότι θα πρέπει ο κόσμος να έχει πράγματι πληροφόρηση, σωστή πληροφόρηση για τα εργαλεία, για τα πάντα κατά την εγγραφή του. Την πρώτη φορά που μοιράζεται πληροφορίες, περιεχόμενο ή χρησιμοποιεί συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του Facebook. Ότι ξέρουν ακριβώς πώς θα προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις για την ιδιωτικότητα στο μέλλον εάν αυτό επιθυμήσουν. Θέλω να πω και το εξής. Πιστεύουμε ότι οι ρυθμίσεις και όλα αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα ανά ηλικία. Οι ρυθμίσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές για τους ανηλίκους, θα εξαλείφονται, θα αποκλείονται αυτομάτως, θα μειώνεται η ορατότητα των ανηλίκων. Δεν θα είναι τα προφίλ των ανηλίκων στις δημόσιες λίστες έρευνας και αναζήτησης επαφών και καθεξής. Εμείς έχουμε προσυπογράψει στην ε, αυτορυθμιστική πρωτοβουλία, ούτως ώστε το διαδίκτυο να είναι καλύτερο και πιο ασφαλές μέρος για τα παιδιά. Και είναι μια πρωτοβουλία που στηρίζει πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε γενικές γραμμές και γενικά μιλώντας, η ιδιωτικότητα από σχεδιασμό by design είναι η σωστή προσέγγιση, δεν ε, ε, δημιουργεί προβλήματα και μπορεί η τεχνολογία να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους χρήστες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα δεν θα υστερήσει, δεν θα καθυστερήσει έναντι των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και θα λάβουμε υπόψη μας επίσης και όλες τις επιταγές και προσταγές ως προς την ιδιωτική σφαίρα και την ιδιωτικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε Έρικα για την ομιλία σου. Και τώρα είναι μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω τον επόμενο ομιλητή μας, τον κύριο Αλεξάνδρ Ντίξ υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων και την ελευθερία τη ε, πληροφόρηση στο Βερολίνο στη Γερμανία. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Αχή για αυτή την ευγενική παρουσίαση. Είναι τιμή μου να μπορώ να απευθυνθώ στου βουλευτέ του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχω δέκα σημεία και μια τελική παρατήρηση που θα ήθελα να σα υποβάλω. Καταρχάς, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν κανονισμό ε, προστασίας, για ένα γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, έχει στόχο να διασφαλίσει ένα νομισμένο υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ωστόσο, όπως ε, η Οδηγία 9546 δηλώνει στην αιτιολογική σκέψη 10, η προσέγγιση των νόμων των κατώμελών μελών δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της προστασίας που ήδη προσφέρεται. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για την εναρμόνιση που προκύπτει από την εφαρμογή κανονισμού και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, να δηλωθεί σαφώς το κείμενο του κανονισμού. Ένα παράδειγμα που ήδη αναφέρθηκε από προηγούμενους ομιλητές η περισσότερη ευελιξία χρειάζεται για τα κατημέλη σε ορισμένους ειδικά τομείς, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης ειδικά σε αυτό το τομέα, όχι μόνο σε αυτόν. Το άρθρο 82 ε, του σχεδίου κανονισμού είναι ιδιαίτερα ε, περιορισμένο και ιδιαίτερα σαφές κατά την άποψή μου. Διότι τα κάτι μελη έχουν τη δυνατότητα να νομοθετήσουν στον τομέα της απασχόλησης μόνον εντός των ορίων του κανονισμού. Στη Γερμανία, όπως το αναφέρει και ο Στέφαν Μάγερ, υπάρχουν νόμοι και συμφωνίες που επιτρέπουν ε, συγκεκριμένη προστασία των εργαζομένων και των όσων υποβάλλουν αίτηση αναζητούν εργασία. Αλλά δεν είναι σαφές εάν μέσω του κανονισμού, εάν θα ισχύουν ε, οι κανονισμοί και οι συμφωνίες και μετά την έγκριση του ευρωπαϊκού κανονισμού. Οι ευρωπαϊκοί νομοθέτες δεν πρέπει να υποβαθμίσουν το επίπεδο προστασία για την εναρμόνιση, επειδή θα πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο προστασία και όχι να γίνει ένα αγώνα δρόμου προ την υποβάθμιση. Σωστά είπε και ο κ. Σούλς το πρωί ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μέσος όρος επαρκούς προστασίας και αυτό θα πρέπει να προκύπτει από το 82 εφόσον διευκρινιστεί. Τώρα για τις ειδικέ διατάξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να λάβει ειδικέ προβλέψεις ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως νομίζω ότι ο αριθμός και ο βαθμός των εξαιρέσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι υπερβολικός. Ένα παράδειγμα για την προστασία των παιδιών. Εάν συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρξουν ειδικέ διατάξει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ενό παιδιού, δεν καταλαβαίνω να μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση κάποια μικρομεσαία επιχείρηση να συζητιέται εάν χρειάζεται την ε, παλιθευόμενη συγκατάθεση ή όχι βάσει του άρθρου 8. Ε, το όριο των 250 εργαζομένων για τον ορισμό υπευθύνου της επεξεργασίας δεδομένων μου φαίνεται παράλογο, διότι θα μπορούσε μια χαλιβουργία που έχει 250 εργαζομένους ε, στον τομέα τη επεξεργασία του Χάλιβα να έχει και δύο υπαλλήλου για την επεξεργασία των δεδομένων. Είναι θέμα υποχρέωση, Ε, αλλά κάποιοι άλλοι γιατροί, λόγου χάρη, με πέντε υπαλλήλου που χειρίζονται τόσο ευαίσθητα δεδομένα αυτά το, που αφορούν την υγεία των ε, πολιτών μα, δεν θα έχουν τέτοια υποχρέωση για υπευθύνου επεξεργασία δεδομένων. Τώρα, ο ορισμό του έλεγκτη και του υπευθύνου τη επεξεργασία ο κανονισμός φαίνεται ότι έχει αντλήσει διδάγματα από την περίπτωση του SWIFT και το άρθρο 24 μιλά για την κοινή εποπτεία. Όμως τα άρθρα 82 και 88 είναι κάπως ασαφή ο διαχωρισμός μεταξύ του ελεγκτή και του υπευθύνου επεξεργασίας. Ορίζονται για τον ελεγκτή στο 22, ενώ στο 28 αναφέρεται η τεκμηρίωση και για τους ελεγκτές και για τους υπευθύνους επεξεργασίας, για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας. και αναφέρονται και οι ευθύνε με τον ισχύοντα νόμο. Ο υπεύθυνο τη επεξεργασία νομικό αποτελεί μέρο των αρμοδιοτήτων του ελεγκτή. Οπότε δεν έχει δικέ του ανεξάρτητε αρμοδιότητε, έχει καθήκοντα αλλά εδώ φαίνεται να είναι ατυχής η διατύπωση του κειμένου. Θα χρειαστεί λοιπόν διευκρίνηση, διότι αυτό που απαιτείται είναι η ευθύνη να μην εξατμιστεί στο συσχετισμό της εργασίας των ελεγκτών με του ε, ε, υπευθύνου επεξεργασία, στην περίπτωση λόγου χάρη του υπολογιστικού νέφους. Τώρα για την ε, αγορα, για την εμπορία θα πρέπει εδώ να υπάρχει η συνειδητή συγκατάθεση ή λόγου χάρη η εντολή do not track ως αυτόματη ρύθμιση. Αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένη νομική βάση, όπως το άρθρο 6.1 από το Β ως το ΣΥΓΜΑΤΑ. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το άρθρο 19.2 και η ιδεολογική σκέψη 57 να εξελιχθούν πλήρως. Θα πρέπει τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα σε όλους αυτούς τους τομείς. Έπειτα, θα πρέπει να προβλεφθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείται ψευδόνυμο για τα προσωπικό δεδομένα των ε, πολιτών, των ατόμων. Και αυτό θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία του ιδιωτικού βίου βάσει σχεδιασμού. Έπειτα, ο συσχετισμό μεταξύ του κανονισμού και τη οδηγία για την ηλεκτρονικό ιδιωτικό βίο. Το άρθρο 89 εγείρει περισσότερα ερωτήματα από ό,τι καλύπτει απορίε. Η ε, ανεπαρκή διάκριση μεταξύ του γενικότερου πλαισίου και τη συγκεκριμένη δευτερογενή νομοθεσία προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πρόβλημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποιε από τι διατάξει του σχεδίου κανονισμού όντω κοιτάζουν ορισμένα ζητήματα, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο. Ενώ από την άλλη η οδηγία έχει σχεδιαστεί με τρόπο ασαφή κατά την άποψή μου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει βελτίωση. Σίγουρα υπάρχει καλύτερο τρόπο, είτε να ενσωματώσουμε του κανόνε προστασία δεδομένων για τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Συνολικά είναι τεράστιο έργο, αλλά θα πρέπει να το φέρουμε ει πέρα, είτε να γίνει καλύτερη διάκριση μέσω τη ανάλογη διάταξη. Έβδομη παρατήρηση, και αυτό το ανέφερε και η Ισπανίδα εκπρόσωπο νωρίτερα, η σχέση μεταξύ του κανονισμού και τη οδηγία από τη μια και των νόμων για την ελευθερία τη πληροφόρηση στα κράτη-μέλη. Ο ζητημό αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Προ στιγμή, αυτό γίνεται μόνο σε μία αιτιολογική σκέψη. Εγώ θα ήμουν ε, υπέρ μιας ε, πολύ συγκεκριμένης διάταξης, έστω γενικού χαρακτήρα, αλλά στο ίδιο το κείμενο του κανονισμού και της οδηγίας, που να μην αφορά μόνο το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί όλο ένα και περισσότερα κάτι μέλη προβλέπουν υποχρεώσεις διαφάνειας και πρόσβαση στην πληροφορία. Εδώ η πρόταση θα ε, είναι ολοκληρωμένη όταν φτάσουμε σε μια ε, τέτοια διευκρίνηση, με μια διάταξη που να εξηγεί αυτόν τον συσχετισμό. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ μια τέτοια διευκρίνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ανέφερα και προηγουμένω, ε, προποθέτει ότι το σχέδιο κανονισμού θα. Ε, υπερισχύει. Βεβαίω, η καταξιοδότηση πράξη είναι κάτι που κυρίω θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω και τον έλεγχο μέσω του μηχανισμού συνεκτικότητα. Όμω, οι ευρωπαϊκοί νομοθέτε θα πρέπει να μπορούν να, καθαρίσουν, να καθορίσουν ε, τα κέρια σημεία του κανονισμού, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι, πράξει μπορούν να εγκριθούν, αλλά και η ομάδα εργασίας του 29 μόλις ενέκρινε ένα διεξοδικό έγγραφο εργασίας, όπου αναλύει και μελετά τις διατάξεις που οδηγούν στην έγκριση πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Κάνει και συγκεκριμένε πρακτικέ συστάσει για το πώ να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Σα παραπέμπω στο σχετικό έγγραφο εργασία. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μηχανισμό ελέγχου συνεκτικότητα, δεν συνάδει με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ανεξαρτησία των ε, αρχών επίβλεψη. Η ένατη παρατήρησή μου έχει να κάνει με την ενιαία θηρίδα, δηλαδή τι διατάξει περί μονοπευθυντική θηρίδα. Νομίζω η φιλοσοφία αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνον εφόσον είναι ηγετικό ρόλο τη φορέα αυτού τη ενία θηρίδα. Θα πρέπει όμω και τα κράτη-μέλη να μπορούν να ενημερώνουν τι νομικέ αρχέ για του συγκεκριμένου εθνικού του κανόνε για την προστασία των δεδομένων που δεν έχουν εναρμονιστεί. Α είμαστε ρεαλιστέ και ειλικρινεί. Το σχέδιο κανονισμού δεν θα πετύχει την πλήρη εναρμόνιση, δεν θα γίνει εναρμόνιση 100%. Πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι τομεί, όπω το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, άλλοι τομεί, που θα υπάρχουν ειδικέ διατάξει για την προστασία των δεδομένων και θα πρέπει οι εθνικοί ελεγκτέ, οι εθνικέ αρχέ δηλαδή, να μπορούν να επηρεάσουν τόσο προτείνει η αρχή που έχει ηγετικό ρόλο. Αυτό δεν τα επιλύει, δεν τα επιλύει ο μηχανισμό συνεκτικότητα. Δέκατη παρατήρηση, ο ρόλος των αρχών επίβλεψης ε, και των ανάλογων φορέων. Το άρθρο 24 για την παρακολούθηση θα οδηγήσει σε αύξηση του φόρτου των σημερινών ε, ε, εθνικών υπευθύνων που έχουν ήδη περιορισμένους πόρους στα περισσότερα κάτι μέλη. Η κατάσταση αυτή πραγματικά θα ε, επιταθεί εφόσον εγκριθεί το 24 και δεν προσαρμοστεί. Θα πρέπει να μπορεί να προσφύγει με ένδικα μέσα ο πολίτης για τον οποίο έχουν συλλέγει τα δεδομένα, εφόσον θέλει να μηνύσει, ας πούμε, τον ε, επιθεωρητή των ε, προσωπικών δεδομένων ή να μηνύσει τον ε, υπεύθυνο κάποια άλλη χώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή είναι η να μηνυσει τον υπευθυνο καποιες αλλες χωρα εγω προσέγγιση. Οι σφραγίδε και τα σήματα είναι η καταλληλότερη λύση και αυτό θα μπορούσε να μας το παράσει και το άρθρο 29. Τελευταία παρατήρηση. Παρόλο που το σχέδιο κανονισμού είναι τεχνολογικός ουδέτερο στι εκφράσεις του, ήταν πολύ καλή η πρόταση του καθηγητά, καθηγητή κυρίου Σιμίτη. Θα πρέπει να υπάρχει και μία ρήτρα sunset με βαθμιαία ε, αναθεώρηση. Δεν μπορεί να παραμείνει ο κανονισμός αυτός απαράλλακτος για 20-30 χρόνια. Σοβαρά πρέπει να σκεφτούμε ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή όχι απλώς αποτίμηση, αλλά ίσως και μια ρητρα sunset με βαθμιαια αναθεωρηση δεν μπορει να παραμεινει ο κανονισμος αυτος απαραλλακτος για 20 30 χρονια σοβαρα πρεπει να σκεφτουμε οτι θα χρειαστει καποια στιγμη οχι απλως αποτιμηση αλλα ισως και μια ρητρα sunset. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστώ, Αλεξάνδερ. Μιλήσαμε για το Facebook, μιλήσαμε για το ρήτρα Σάρσετ. Τώρα να περάσουμε στον ιδιωτικό, βάση, ε, ιδιωτικό βίο βάση σχεδιασμού, την προστασία της ιδιωτικότητας βάση σχεδιασμού και να ακούσουμε τον κύριο Αρμίν Τουτίν που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχετε το λόγο κύριε Τουτίν. thank you very much. Uh, I will speak in... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Έχω προετοιμάσει και κάποιε διαφάνειε. Ε, Δυστυχώ δεν μπόρεσα να τι ετοιμάσω στα αγγλικά γιατί δεν είχα αρκετό χρόνο για να τα μεταφράσω. Τα έγραψα στα, στα γερμανικά και θα κάνω και την παρουσίασή μου στα γερμανικά. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα μιλήσω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπου είμαι μέλο τη ομάδα μελέτη για τον κανονισμό δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΕΟΚΕ για την οδηγία και δεν υπήρχε ομάδα μελέτης ε, για την οδηγία. Αλλά εμείς περισσότερο ε, λαμβάνουμε το λόγο από την πλευρά των εργαζομένων και πολλά από τα σημεία που αναφέρονται σε αυτές τις διαφάνειες είναι σημεία που συζητήθηκαν από την ΕΟΚΕ και θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες. Πολλά σημεία έχουν ήδη αναφερθεί από πολλούς προλαλήσαντες ομιλητές, από τον κύριο Ντίξ παραδείγματος χάρη. Ένα σημείο δεν έχει αναφερθεί όμως ακόμη, ή τουλάχιστον δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς. Από την πλευρά των εργαζομένων θεωρούμε ότι το θέμα της προστασίας των δεδομένων πρέπει να έχει το προβάδισμα, σαφές προβάδισμα έναντι άλλων στοιχείων όπως είναι οι ελευθερίες στην ε, ε, εσωτερική αγορά. Υπάρχει η οδηγία του 95 και βρίσκονται και τα δύο αγαθά σε ίδιο επίπεδο, δηλαδή η προστασία των δεδομένων και η ελευθερία στην εσωτερική αγορά. Θα έπρεπε να έχει το προβάδισμα ε, η προστασία των δεδομένων, το θεμελιώδες ε, δικαίωμα για την προστασία δεδομένων και υπάρχει το δικαίωμα αυτοδιαχείρισης όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Στην Γερμανία είναι πολύ ε, υψηλή η αξία της προστασίας δεδομένων. Στη γνωμοδότησή της η ΕΟΚΕ λέγει ότι η επεξεργασία και μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της ενιαίας αγορά θα πρέπει να περιορίζεται από το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά του, ε, της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων και εδώ υπάρχει το Συνδικάτο Βέρντι ε, εκπροσωπείται στο Σύνδεσμο Γερμανικών Συνδικάτων και εγώ δουλεύω για το Συνδικάτο Βέρντι ε, και λέμε ότι θα πρέπει το το μέσο το οποίο προτείνεται, το οποίο προτείνεται είναι ένας κανονισμός, πρέπει να δούμε ποια στοιχεία ε, περιλαμβάνει ως κανονισμός. Τα ανέφερε και ο κύριος Μάγερ και ο κύριος Ντίξ και πρέπει να δούμε αν ε, και σε εθνικό επίπεδο αυτά τα οποία υπάρχουν θα παραμείνουν σε ισχύ ή θα πρέπει να δούμε και τι ρόλο παίζει το άρθρο 82 σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βλέπουμε ότι δεν ε, πρέπει ε, να παρεκκλίνουμε από τα υψηλά πρότυπα. Ένα πρόβλημα είναι το σε ποιο δικαστήριο θα στραφεί ένας πολίτης όταν ε, το μέσο το οποίο έχουμε, το νομικό μέσο είναι κανονισμός, θα πρέπει κανείς να στραφεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο και τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια. Και επαναλαμβάνω ότι το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο έχει πάρα πολύ υψηλό ρόλο και έχει θέσει πολύ υψηλέ προδιαγραφέ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήταν ε, το σωστό νομικό μέσο μια οδηγία αντί ενός κανονισμού ούτως ώστε να έχουμε την απαιτούμενη εναρμόνιση. Ε, αυτό είναι θέμα ε, του Ευρωπαίου Νομοθέτητο, πώς θα χειριστούν αυτό το θέμα ε, και πρέπει να δούμε τη διατύπωση του άρθρου 82, όπου λέει στο πλαίσιο του κανονισμού, στο πλαίσιο των ορίων του κανονισμού. Το είπε και ο κύριος Ντίξ αυτό. Η ΕΟΚΕ προτείνει εδώ να λέμε βάση του κανονισμού και όχι ε, στο πλαίσιο του κανονισμού. Για να μπορούμε να έχουμε ε, δυνατότητα παρέκκλησης από τον κανονισμό για να επιτύχουμε υψηλότερα όρια προστασίας δεδομένων. Και αυτό μας ενδιαφέρει και για το άρθρο 80 και τα, επόμενα άρθρα που αφορούν ε, τα δεδομένα ε, στον τομέα της υγείας και τα κοινωνικά δεδομένα. Υπάρχει μια ειδική διάταξη για τη συγκατάθεση και εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Μάγερ. Συμφωνούμε σε πολλά σημεία αλλά όχι σε αυτό. Κατά τη γνώμη μας είναι πολύ καλή η πρόταση της Επιτροπής εδώ για τις αιτιολογικές σκέψεις 25 και 34 και στο άρθρο 7 ε, διότι ε, για τους εργαζομένους ε, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ισότιμη σχέση αλλά υπάρχει σχέση εξάρτησης. Επομένως δεν μπορεί να δίδουν τη συγκατάθεσή τους για την παροχή δεδομένων εφόσον τη δίδουν σε κάποιον από τον οποίο εξαρτώνται. Δεν τίθεται λοιπόν εδώ θέμα συγκατάθεσης. Υπάρχουν ε, προτάσεις που δείχνουν ότι ε, οικειοθελώς παρέχονται αυτά τα δεδομένα και φοβούμαι ότι στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου η συζήτηση που γίνεται ε, μειώνει το θετικό χαρακτήρα της πρότασης της Επιτροπής και θα ήθελα εγώ να παραμείνει η πρόταση της Επιτροπής ως έχει στο άρθρο 7 για να μην μειωθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Το θέμα τώρα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε μια επιχείρηση προτείνεται ένα κατόφλι των 250 εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι το 60% των απασχολουμένων, το 60% των εργαζομένων μένουν εκτός του τομέα προστασίας. Το υπολογίσαμε με βάση στατιστικά δεδομένα της Eurostat για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στη Γερμανία αυτό θα είχε ως συνέπεια το 90% των εργαζομένων ε, που εργάζονται σε επιχειρήσεις που μέχρι τώρα θα είχαν υπεύθυνο προστασία δεδομένων, στο εξή δεν θα έχουν με αυτές τις διατάξεις. Και αυτό δεν μπορεί να, γίνει αποδεκτό. Η ανεξαρτησία του υπεύθυνου προστασία δεδομένων πρέπει να είναι εγγυημένη και αναφέρουμε διάφορες ε, απαιτήσεις, την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης, την προστασία ε, από απόλυση. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε Συμβούλια Επιχειρήσεων να προστατεύονται και μετά τη θητεία τους ε, σε τέτοια, σε τέτοια όργανα. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κατάρτιση για τα νομικά θέματα και να μην υπάρχει υποχρέωση κοινοποίηση των παραβάσεων στους εργοδότες και να υπάρχει απαλλαγή από την ευθύνη. Το κατόφλι θα πρέπει να μειωθεί στα 20 άτομα, δηλαδή τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την συλλογή δεδομένων και την επεξεργασία τους ε, και τα όρια τα οποία, ε, ή αν δεν, ισχύσουν, δεν ισχύσει αυτό το όριο των 20 ατόμων για την προστασία των, που ισχύσει η Γερμανία για την προστασία των δεδομένων, θα πρέπει να ισχύσουν τα όρια που ισχύουν για τη δημιουργία συμβουλίων ε, εκπροσώπησης εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Άλλες κατηγορίες όπως δεδομένα για την ε, υγεία ή κοινωνικά δεδομένα. Εδώ υπάρχουν διάφορα κενά στην νομοθεσία. και θα πρέπει ε, να απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων για το αν ανήκουν οι εργαζόμενοι σε συνδικάτα, να μην συμπεριλαμβάνονται δεδομένα ε, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, να μην υπάρχουν ε, επίσης δεδομένα τα οποία παρανόμως έχουν ε, αποκτηθεί και να μην υπάρχουν στοιχεία από τεστ προσωπικότητας ή ερωτηματολόγια προς τους εργαζομένους, ούτε γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα. Νομίζω ότι έχω ξεπεράσει τον χρόνο μου και θα προσπαθήσω να συντομεύω. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μας είναι τα δικαιώματα ε, της εκπροσώπησης ε, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Η αρχή της μονοαπευθυντικής θηρίδας δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο ότι δεν θα μπορούν να παίξουν το ρόλο τους επιτόπου οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων ή οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην επιχείρηση. ο ευρωπαϊκός κανονισμός θα πρέπει να θέτει πολύ υψηλά πρότυπα, αλλά φοβόμαστε ότι δεν θα είναι τόσο υψηλά τα πρότυπα ε, όσο είναι σε ορισμένα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρχουν αυτά τα μέτρα διασφάλισης. Και όταν υπάρχουν διασυνοριακές ανταλλαγές δεδομένων, πάλι θα πρέπει να παίζουν το ρόλο ε, οι υπεύθυνοι δεδομένων στις επιχειρήσεις. Ανέφερε και ο κύριος Μάγερ το θέμα της, ε, των συλλογικών αγωγών, εκ μέρους σωματείων παραδείγματο χάρη, οι οργανώσεις καταναλωτών οι οργανώσει καταναλωτών κάνουν συλλογικέ αγωγέ για του καταναλωτέ και θα πρέπει του εργαζομένου να μπορούν να του εκπροσωπούν τα συνδικάτα του ή τα αναγνωρισμένα ε, συλλογικά του όργανα. Αναφέρθηκε και το θέμα των πράξεων κατεξουσιοδότηση. Ε, και δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Θα μιλήσω όμως για τα προνόμια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, θα διαφωνήσω με κάποιους από τους προλαλήσαντες. Δεν βλέπουμε γιατί θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια διάκριση μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονται σε μικρές ε, επιχειρήσεις ε, με λιγότερους από 250 ή με περισσότερους από 250 εργαζομένους. Το ότι εργάζεται κάποιος σε μία μικρή επιχείρηση δεν θα πρέπει να οδηγεί στο ότι δεν θα υπάρχει προστασία των προσωπικών του δεδομένων και θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται. Και ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα πρέπει ε, να θεσπίσει τους κατάλληλους κανόνες και να διορθώσει σε αυτό το σημείο την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μποργέζιους από το Ινστιτούτο Δικαίου πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Σα παρακαλώ όμω να κρατήσετε το χρόνο των 10 λεπτών γιατί μέχρι τι 6 ε, και 45 μπορούμε να έχουμε διερμηνία, αλλά όχι αργότερα. Και επειδή θέλουμε να έχουμε ερωτήσει από το ακροατήριο με διερμηνία, παρακαλώ μην υπερβείτε το χρόνο σα. Καλησπέρα σα κύριε και κύριοι. Έχει περάσει η ώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν ε, να παραμείνω σε μια ελαφρά παρουσίαση με δύο σημεία. Η μία είναι τεχνικού χαρακτήρα και το επόμενο είναι ακόμη πιο εύκολο. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Θα έπρεπε νομίζω ο ορισμός όχι των προσωπικών δεδομένων, αλλά του υποκειμένου των δεδομένων να τροποποιηθεί, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα ε, για να απομονωθεί, να κατομικευθεί κάποιος. Ε, αυτό θα πρέπει να υπάρχει στον ορισμό για να μην μπορεί μια επιχείρηση να εντοπίσει κάποιον ακόμη και αν δεν έχει το όνομά του και έπειτα θα πρέπει να διευκρινιστούν οι διατάξεις που αφορούν την συγκατάθεση στον, ε, στην πρόταση κανονισμού. Για το πρώτο λοιπόν σημείο. Ο ορισμός των ε, προσωπικών δεδομένων είναι ο πιο σημαντικός ολόκληρου του κανονισμού. Διότι αν δεν ορίσουμε τι είναι πρόσωπο, δεν ορίζονται και τα προσωπικά δεδομένα και δεν ισχύει ο κανονισμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε στη διαφάνεια. Αυτό που γράφει το κείμενο είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξατομικευθεί κάποιος ή να ε, ξεχωριστεί μέσα σε μια ομάδα. Αυτά θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η ορθή ερμηνεία της ισχύουσας οδηγίας, αλλά το λέμε εδώ και πέντε χρόνια. Σταθερά ότι δεν υπάρχει ανώτατο δικαστήριο που να έχει καλύψει κάτι τέτοιο με την ομολογία του. Καλό λοιπόν θα είναι να δοθεί έμφαση στον κανονισμό είναι μια νέα, δεν είναι μια νέα διάσταση, γι' αυτό ακριβώ πρέπει να δοθεί έμφαση. Γιατί κάνω αυτή την τεχνική παρατήρηση. Να σα δώσω ένα-δύο παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο σκόπιμο θα είναι αυτό στην πράξη. Πολλέ δραστηριότητε επεξεργασία των δεδομένων σήμερα, ιδίω στο διαδίκτυο, έχουν τρομέρε λεπτομέρειε για προσωπικά προφίλ, Τρομερέ λεπτομέρειε. Όμω οι εταιρείε μπορεί να μην θέλουν ή να μην χρειάζονται το όνομα του κατόχου των δεδομένων. Μπορεί όμω να έχουν λεπτομερέστατα προφίλ στα χέρια του, τα οποία πριν 10-20 χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμπεριφορά ε, από τι διαφημιστικές εταιρείε. Μπορεί να ερευνήσουν τη συμπεριφορά των προσώπων ή ακόμη και μέσω του Twitter με ένα ψευδόνυμο να αντλήσουν στοιχεία. Μπορούν λοιπόν να παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάποιου, τα cookies ή με τον εντοπισμό μιας συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εντοπισμού μέσω ενός smartphone και αυτά σήμερα μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένα τεχνολογικώς αλλά σε 10 χρόνια θα υπάρχουν. Τα προφίλ λοιπόν αυτά μπορούν να είναι λεπτομερέστατα και θα θυμάμαι χθε μόλις ε, συνάντησα εκπροσώπους μιας διαφημιστικής εταιρείας ε, οι οποίοι είχαν 70.000 στοιχεία αναπροφίλ, αλλά η εταιρεία λέει ότι δεν μπορεί να αποδώσει ονόματα στα συγκεκριμένα προφίλ. Δεν λέω να απαγορευτούν αυτέ οι επιχειρηματικέ πρακτικέ, όμω αν αυτά τα προφίλ θέλουμε να μείνουν εκτό του κανονισμού, τότε είναι σαν να μην έχει νόημα ο κανονισμό. Εάν τα προφίλ αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό, τουλάχιστον θα υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει για τη συγκατάθεση, τη διαφάνεια και το καθεξής. Η διαφάνεια ε, περιλαμβάνει μια εικόνα για τις εταιρείε που μελετούν την συμπεριφορά. Ένα παράδειγμα ενός ανώνυμου προφίλ εντός ε, εισαγωγικών ή τέλος πάντων με ψευδόνυμο. Βλέπετε, για το άτομο αυτό ξέρουν την ηλικία του, ξέρουν ότι έχει δύο παιδιά, ξέρουν ε, σε το ταχυδρομικό του κώδικα. Ξέρουν ότι κερδίζει περίπου 150 έως 160 χιλιάδες δολάρια Και ούτω καθεξής. Το μόνο που τους λείπει ή το ε, έσβησαν μόνοι τους είναι το όνομα. Αυτή λοιπόν η απεικόνηση, αυτή η περίπτωση θεωρώ ότι μπορεί να καλύπτεται από τον κανονισμό. Ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς ένα ανώνυμο προφίλ ε, μπορεί να μοιάζει. Φανταστείτε, μια εταιρεία marketing, αυτό σημαίνει συχνότητα, που μέσα από ένα smartphone ε, μπορεί να εντοπίσει μια τοποθεσία. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα με όλα τα smartphone, αλλά σε κάποια χρόνια μπορεί να είναι περισσότερα τα προϊόντα που έχουν δυνατότητε εντοπισμού με GPS. Μπορεί κάποιο λοιπόν να μπορεί να ε, εντοπίσει κάποιον μέσω της τοποθεσίας και όχι αναγκαστικά μέσω του ονόματος και να χρησιμοποιήσει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά. 70.000 ε, στοιχεία, χαρακτηριστικά λοιπόν αναπροφίλ μπορεί να έχει η εταιρεία, θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να ισχύει ο κανονισμός. Ε, ε, τονίζω ότι δεν πρόκειται για απαιτήσει απαγόρευση εδώ. Όχι. Απλώ θα πρέπει να καλύπτονται αυτοί οι κανόνε, ε, να καλύπτουν οι κανόνε και τη μελέτη τη συμπεριφορά τη προσωπικότητα. Αυτό είναι σχεδόν ε, το τέλος της πρώτης μου παρατήρησης. Μια μικρή λεπτομέρεια που θα πρέπει να την αναφέρουμε ξεχωριστά. Η τηλογική σκέψη 24 περιγράφει τα είδη προφίλ που μόλις σας παρουσίασα. Το, η τηλογική σκέψη 24 λέει λίγο πολύ ότι τα άτομα μπορεί να εντοπιστούν με συγκεκριμένα στοιχεία όπως τα κούκκις και μπορεί να μείνουν ίχνη τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε τελικά να διαμορφωθεί το προφίλ τους. Συμφωνώ απολύτως με αυτό, αλλά προτείνω τελευταία πρόταση να διαγραφεί. Η τελευταία πρόταση προκαλεί σύγχυση. Προσθέθηκε μάλιστα λίγες εβδομάδες μόλις πριν την ε, δημοσιοποίηση της τωρινής πρότασης. Είναι συγκεχημένη η διατύπωση και η τελευταία πρόταση δίνει μια συγκεκριμένη χρειάστη διατύπωση, αλλά καλό θα ήταν να διαγραφεί. Αυτό ήταν το τεχνικότερο ζήτημα που ήθελα να αναπτύξω. Τώρα, οι πληροφορίε που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να εντοπιστεί κάποιο, να εξατομικευθεί κάποιο, θα πρέπει να εμπίπτουν στο τοπικό του κανονισμό. Αυτό δεν είναι τίποτα το επαναστατικό. Το άρθρο 29 εν μέρη το αναφέρει και πολλοί το λένε εδώ και χρόνια. Το δεύτερο είναι πολύ απλό. Παρακαλώ μην μειώσετε τις απαιτήσει για τη συγκατάθεση. Δεν πρέπει, μάλλον θα πρέπει η συγκατάθεση να είναι και συνειδητή και τεκμηριωμένη και να δίνεται ελεύθερα. Θα πρέπει να είναι ένδειξη της βούληση κάποιου. Αυτό είναι πολύ λογικό. Όμως κάποιοι επισημαίνουν ότι η πλήρης σιωπή ή η αδράνεια συχνά ερμηνεύεται ως συγκατάθεση. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι γενικώ έτσι θα πρέπει να ε, αντλείται η συγκατάθεση. Αυτό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει μέσω της πρότασης και καλό θα πρεπει να ισχυει μεσω τη προταση και καλο θα ειναι να το φροντίσουμε. Εάν οι προδιαγραφέ μείνουν ω έχουν, θα μπορούσε να υπάρχει ένα κουτάκι στο κάτω μέρος μιας σελίδα σε έναν ιστότοπο που να λέει ότι εφόσον ε, τσεκάρει κανείς αυτό το κουτάκι έχει δεχτεί τη δυνατότητα αλλαγής των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν την ε, χρήση του στο Λοιπόν, αυτό δεν θα πρέπει να μπορεί να επιτραπεί. Δεν θα πρέπει να υποβαθμίσουμε τις απαιτήσει, αλλά να μείνουν ως έχουν. Ορθώς το τονίζει το εκτιμώντας 26. Λέει λίγο πολύ ότι η σιωπή ή η αδράνεια δεν αποτελούν συγκατάθεση. Παρακαλώ αυτό να ισχύσει. Έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Ε, ανακεφαλαιώνοντας, η πρώτη παρατήρηση νομίζω ήταν κάπως περιπλοκότερη, πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε κανείς να εξατομικεύεται ή τέλος πάντων να παρακολουθείτε ή να στοχοποιείτε. Αυτά ούτως ή άλλως στο πεδίο ορισμού υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν. Είναι και στο πεδίο του κανονισμού. Η δεύτερη παρατήρηση παρακαλώ μην χαμηλώσετε τον πύχη για την συγκατάθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εάν δεν έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τώρα, εδώ, ευχαρίστως να απαντήσω στις ερωτήσεις σας μέσω mail. Ε, thank you Ευχαριστούμε πολύ, Φρέντερικ. Μας έδωσε στροφή για σκέψη σε όλους. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε όσους ήρθαν να ακούσουν. Το μέλος από τη Γερμανική Βουλή ο κύριος Κωνσταντίν Βον Νότς. Δύο λεπτά. Το ανώτατο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλε τι παρεμβάσει που ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Θα είμαι σύντομο γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι χαιρετίζουμε το ότι ο κανονισμό αφορά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και νομίζω ότι ε, αυτό είναι ενδιαφέρον ε, ε, και σημαντικό διότι καλύπτουν επιχειρήσεις όπως και το Facebook. Μια ερώτηση και προς τον κύριο Ντίξ θα ήθελα να κάνω. Πώς βλέπετε τον κανονισμό που υπάρχει μέχρι τώρα σχετικά με τη δημιουργία προφίλ και αν βλέπετε να υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης ή ανάγκη βελτίωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα ήθελα να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις μαζί, να μην χάνουμε χρόνο. Πάλι από το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το κύριο Ράχενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι ε, συμφωνώ με αυτό που πολλές φορές αναφέρθηκε στις παρεμβάσει των ομιλητών, ότι ε, δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουμε από τους βασικούς κανόνες προστασίας δεδομένων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ε, χάρη οικονομικών βλέψεων. Και νομίζω ότι ε, στο θεμελιώδες δίκαιο όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει το ότι ε, το δικαίωμα στην ακαιρεότητα του ατόμου και είναι αναπόσπαστα δικαιώματα ε, και προσωπικές θεμελιώδεις ελευθερίες αυτές που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν περισσότερο από ό,τι τα δικαιώματα των επιχειρήσεων στον τομέα των δεδομένων και συγκεκριμένα για τη συλλογή δεδομένων που οδηγούν σε κατάρτιση ενός προφίλ του ατόμου θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το πώς βλέπετε το μέλλον, γιατί πριν από δύο χρόνια μας είχαν πει ότι δεν υπάρχει το θέμα της ε, ταυτοποίησης και αναγνώρισης. Τώρα όμως υπάρχει το personal targeting και το θέμα της ανωνυμοποίησης των δεδομένων ή της χρήσης ψευδονύμου, κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός του αυτός που είναι αντικείμενο της συλλογής δεδομένων στην, στο άρθρο 82 αναφέρονται δεδομένα που αφορούν ε, το εργατικό δίκαιο και ήδη υπάρχουν διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των δικαιωμάτων ε, των εργαζομένων. θα πρέπει να θεσπιστούν τέτοιες διατάξεις που να παρέχουν επαρκή προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιτρέπεται μία παρέκκληση αλλά μόνο προς τα πάνω για αύξηση δηλαδή του βαθμού ε, προστασίας. Θεωρώ ότι αυτή είναι η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μην φυγούν ήδη υπάρχοντα δικαιώματα των προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Περνούμε σε ένα μέλος από την Πολωνική Γερουσία. Μίκελ Σαορνίσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου με τον κύριο Αλεξάνδερ Ντίξ, τον κύριο Ντούτιν, Ρουτίν και τους δύο κυρίους από την Γερμανική Βουλή. Ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει μία διάταξη βάσει της οποίας ε, θα προβλέπεται ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να υπερτερεί εναντί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε πράγματι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο ή τον, το κάθε άτομο που είναι ε, ο ενάγων, ο ενδυνάμει ενάγων. Και είναι αυτή η άποψή μου πραγματικά, διότι είδα αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση το μόνο που κάνουμε είναι να ε, αυξάνουμε τη δουλειά των δικηγόρων. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση των ε, συλλογικών συμβάσεων ή άλλων τέτοιων ε, ρυθμίσεων και εκεί η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να υπερτερεί έναντι των ευρωπαϊκών κανονισμών. Διότι, το λέω αυτό διότι, ο ρόλος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα ε, στο εργασιακό δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο δεν είναι να μειώσει τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά ακριβώς να τα ενισχύσει και να τα προστατεύσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακόμη δύο ζητούν το λόγο. Θα πρέπει όμως να είστε πάρα πολύ σύντομοι γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Η κυρία Μπατέτ από τους Ισπανούς Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρία λόγω του περιεχομένου των παρεμβάσεων και πάρα πολύ χρήσιμη. Ε, έτσι καταλάβαμε ποια είναι η γερμανική θέση η οποία εκπροσωπείται τα μάλλα στο Προεδρείο. Ήθελα να πω τρία πράγματα. Πρώτον, ως προς αυτό το οποίο σχολίασε η κυρία Μαν. Θεωρώ ότι ενδεχομένως εξέφρασε μία δυσφορία ως προς την ιδιωτικότητα λόγω του σχεδιασμού, της δυνατότητας του σχεδιασμού που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία εκπροσωπεί. Αλλά πάντοτε το λογισμικό μπορεί να βελτιωθεί, έτσι δεν είναι. Το εξορισμού by default μπορεί να μην είναι ανοιχτό για όλους, να είναι εξορισμού κλειστό το εξορισμού και να ανοιχτεί μετά από ρητό αίτημα του χρήστη. Υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες, τεχνικά μπορεί να βελτιωθεί το θέμα του, λογιστικού, του λογισμικού. Είναι σημαντικό να έχουν οι χρήστες ένα κλειδί ώστε να έχουν περισσότερη νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου για την ιδιωτική τους ζωή. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερος ο προβληματισμός που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πράγματι, στην Ισπανία το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτό το όριο των 250 εργαζομένων. Άρα το 90% θα αποκλείονταν από αυτό αυτή τη διατύπωση και από αυτή τη διάταξη. Δεν είναι το θέμα μόνο να φτάσουμε στο κατόφλι των εργαζομένων. Το θέμα είναι να συμπεριλάβουμε και τη φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Δηλαδή μια ιδιωτική κλινική μπορεί να έχει πέντε εργαζόμενους μόνο, αλλά να διαχειρίζεται πάρα πολύ ευαίσθητα προσωπικά ε, δεδομένα όπως καταλαβαίνετε. Άρα να τελειοποιήσουμε τα κριτήρια όταν έχουμε να κάνουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η δεύτερη μου παρατήρηση. Και τρίτη παρατήρηση, να εκφράσω την πλήρη μου συμφωνία με τον Φρεντερίκ από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Πράγματι τόνισε τα πιο σημαντικά ζητήματα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα και η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will versuchen, kurz zu Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσετε, παρακαλώ, να είστε ακόμη πιο σύντομοι. Νομίζω ότι σχετικά με αυτό που είπαμε για τη συγκατάθεση είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να είναι όλα προς όφελος των εργοδοτών. Θα πρέπει να αξιολογείται η κατάσταση και βλέπουμε ότι πολλοί ε, εργαζόμενοι ε, φοβούνται να πούν όχι σε μια προσφορά και θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τα δεδομένα από το φόβο να χάσουν την θέση τους σε κάποια προνόμια. Η γραφειοκρατία είναι κάτι το οποίο πρέπει ε, να έχουμε κατά νου και όποτε υπάρχει νέος κανονισμός καταλαβαίνουμε τον επιπλέον άχθος γιατί δεν ε, μιλάμε και για το κόστος και για το διοικητικό άχθος που υπάρχει για τους πολίτες γιατί θα μπορούσε κανείς να ασχολείται μόνο με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Θα έπρεπε και από τους πολίτες να αφαιρεθεί αυτό το βάρος της προστασίας των δεδομένων τους. Όταν είμαι στο Facebook, παραδείγματο χάρη, ή όταν χρησιμοποιώ μια πιστοτική κάρτα, πολύ συχνά ε, αναγκάζομαι να υπογράψω ότι δίνω τα προσωπικά μου δεδομένα και πρέπει κάθε φορά να ασχολούμαι με τεράστιες περιγραφές των ε, στοιχείων τα οποία δίνω κάθε φορά που κάνω κάποια συναλλαγή. Εν πάση δεν θα ακρηγορήσω, είναι αυτονόητα όλα αυτά. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε ε, γραφειοκρατικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις και δεν θέλουμε να αυξάνουμε το κόστος, γιατί και η προσθέση των δεδομένων κοστίζει χρήματα. η προστασία των δεδομένων μπορεί να είναι και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και σήμερα το πρωί το αναφέραμε αυτό, ότι η προστασία των δεδομένων δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε όποτε μπορούμε και όποτε είναι δύσκολο παρετούμε. Θα είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε ακόμη και αν υπάρχει σχετικό κόστος θα πρέπει ε, να μην ε, φιδόμεθα χρημάτων για την προστασία των δεδομένων των πολιτών μας. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσουμε στους συμμετέχοντες στο πάνελ την ευκαιρία να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλες. Σύντομες απαντήσεις παρακαλώ. Από τα αριστερά προς τα δεξιά. Λοιπόν, για την ερώτηση που έχει να κάνει με το μέλλον. Ελπίζω να άκουσα καλά. Εάν δεν άκουσα καλά θα με διορθώσετε. για τα εξανομικευμένα και ενδεχομένως ανώνυμα προφίλ και το τι θα γίνει στο μέλλον. Εάν δεν μιλάμε για τον νόμο, αλλά μιλάμε για την οδηγία, τα προφίλ αυτά νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε καμιά δεκαετία. Εάν λοιπόν μιλάμε για το μέλλον της τεχνολογίας, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό θα απασχολήσει τον τομέα της επεξεργασίας των δεδομένων. Και για το μελλοντικό νόμο, νομίζω πιο εύκολο θα είναι να εφαρμόζεται σωστά ο κανονισμός, εάν προσθεθεί αυτό, αυτό το μικρό κομμάτι, το or singled out, που μπορεί να εξατομικευθεί, να απομονωθεί, να εντοπιστεί. Νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτή τη διατύπωση. Ευχαριστώ. πολύ σύντομα για την παρατήρηση που ακούσαμε από την Πολωνία. Δεν θέλω να με παρανοήσετε. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία για τις εξελαχίστων ε, διατάξεις. Όμως, σε κάποια μέλη σαφώς μπορεί να υπάρχουν καλύτεροι κανόνες. Γι' αυτό δεν θα πρέπει οι καλύτεροι κανόνες να μην μπορούν να ισχύσουν επειδή υπάρχουν οι κοινοτικοί. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε εδώ τους κανόνες, ούτε την εναρμόνιση. Δεν είπα αυτό. Παρακαλώ να με καταλάβετε. Και για να απαντήσω και στην ε, κυρία Μπατέτ, Νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε πάρα πολύ σε αυτό, αλλά σίγουρα η νομοθεσία δεν θα είναι στατική. Η ανταλλαγή δεδομένων θα είναι κάτι το απαραίτητο. Σε κάποιους τομείς θα υπάρχει μεγαλύτερη ανταλλαγή δεδομένων, σε κάποιους άλλους περιορισμένη. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε σοβαρά αυτά. Στην ΕΟΚΕ Ακούστηκαν προτάσεις από την Αυστρία συγκεκριμένα. Μας πρότεινε η Αυστρία κάποιες διατάξεις να χρησιμοποιηθούν για να εκπροσωπηθούν τα συμφέροντα επιχειρήσεων και επίσης να αξιοποιηθούν και για την προστασία των δεδομένων. Απλώς να πω ότι η διερμηνία σταματάει τώρα. Οπότε, εσείς μεταφραστήκατε. Εσείς είσαστε ο τελευταίος που μεταφραστήκατε.